Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε. Το πρώτο θέμα είναι τα πρακτικά. Υπάρχει μια αλλαγή εδώ η οποία έχει προταθεί για την αναβολή του σημείου 17 για το Eurodac με εισηγήτρια την κυρία Μακοβέη πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση του θέματος αυτού. Καλώς ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα πρέπει να επικυρώσουμε τις συστάσεις των συντονιστών για το διορισμό των ακολούθων εισηγητών. Πρώτο, κυρία Μόνικα Μακοβέη για τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βραζιλία για την απαλλαγή θεώρησης για αυτούς οι οποίοι κατέχουν κανονικά διαβατήρια. Δεύτερον, ο, ο συνάδελφος Γιώαν Έντσου για τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Βραζιλία για τους κατόχους διπλωματικών και επισήμων διαβατηρίων. Τρίτον, η κυρία Σίπολ για το δικαίωμα ενημέρωσης για τις ποινικέ διαδικασίες. Και τέταρτον, η κυρία Ρίτα Μπορσελίνο, ιδίας πρωτοβουλίας για τη στρατηγική εσωτερική ασφάλειας. Πόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οι συστάσεις των εισηγητών γίνονται δεκτές. Περνάμε λοιπόν τώρα πριν φτάσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία θα γίνει αργότερα, όπως ζήτησαν ορισμένα μέλη, αντί να περιμένουμε, θα μπορούσαμε να περάσουμε στο σημείο 4. Διεύρυνση της οδηγίας 2003-109 σε αυτούς οι οποίοι την χάνουν διεθνούς προστασίας. Θα ακούσουμε την παρουσίαση της κατάστασης ως έχει σήμερα από τον κύριο Μωράες, ο οποίος θα μας ανημερώσει για τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου που οργανώθηκε για το συγκεκριμένο θέμα να μην ξεχνάμε ότι ένας δεύτερος τριμερής ε, διάλογος προβλέπεται για τις 9 Νοεμβρίου που θα μπορούσε ίσως να είναι ο τελευταίος. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου. Κλόντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα να σας ενημερώσω για τον πρώτο τριμερή διάλογο. Η συνάντηση ήταν επικοδομητική. Ευχαριστώ και τις κοιόδους εισηγητές και εισηγήτριες. Το Συμβούλιο συμφώνησε με τις δικές μας τροπολογίες και στις υπόλοιπες που υπήρχε θέμα καταλήξαμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γι' αυτό. Υπάρχουν όμως κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες θα συζητήσουμε αύριο στα πλαίσια των σκιωδών εισηγητών και στα πλαίσια του επομένου τριμερούς διαλόγου στις 10 Νοεμβρίου. Αφορούν τη χρονική διάρκεια κάλυψης, εδώ το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν ξεκάθαρες απόψεις. Θα τα συζητήσω τα θέματα αυτά με τους σκιώδεις αύριο. Άλλα θέματα σε εκκρεμότητα αφορούν τις απελάσεις μελών οικογενείας, τον μηχανισμό διαβούλευσης σε περίπτωση απέλασης και τις κοινέ αναλήψεις υποχρεώσεων κρατών μελών. Όλα τα θέματα αυτά νομίζω θα επιληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω να υπάρξει λοιπόν σε δύο-τρεις εβδομάδες μια συμφωνία στα πλαίσια του δευτέρου τριμερούς διαλόγου Ελπίζω να φτάσουμε ε, στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο αφού ψηφίσουμε τέλος Νοεμβρίου. Πάντως ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, εισηγητές, κοιόδης και τους συναδέλφους της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την προθυμία που επέδειξαν στη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ Κλοντ για την παρουσίαση. Έχουμε εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου εδώ. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θα ήθελε κάτι να πει. Όχι. Η Προεδρία θα ήθελε κάτι να πει, κάποιο μέλος θα ήθελε κάτι να πει. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ. Α, βλέπω, ναι. Κυρία Νεντέλτσεβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μωράες. Το επαναλαμβάνω, έχει κάνει όμως εξαιρετική δουλειά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι λέγοντας ότι ο τριμερής διάλογος ήταν αρκετά παραγωγικός και πρέπει να βρούμε τώρα λύσεις στις εκκρεμότητες αποδεκτές και για μας και για την Επιτροπή. Τρία σημεία. Καταρχάς το θέμα της ενσωμάτωσης είπαμε ότι τα θέματα των μαθημάτων γλώσσας είναι πολύ ευαίσθητα. Θα ήθελα να υποστηρίξω την θέση που λέει ότι τα μαθήματα γλώσσας είναι στη βάση μιας επιτυχημένης διαδικασίας ενσωμάτωσης. Η αποτυχία των πολιτικών ενσωμάτωσης είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σαφώς και γι' αυτό ακριβώς θα υποστηρίξω την τροπολογία για τα γλωσσικά μαθήματα, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τη θέση του Συμβουλίου που επιμένει στη μορφή των μαθημάτων και στο περιεχόμενο. Για την αποκατάσταση της οικογενειακής ενότητας η συμβιβαστική πρόταση του Συμβουλίου είναι αποδεκτή το τρίτο θέμα για τον μηχανισμό διαβούλευσης ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση κατά την οποία το δεύτερο κράτος μέλος θέλει να προχωρήσει στην απέλαση ενός κατοίκου με μόνιμη κάρτα παραμονής, κατανοώ τις δυσκολίες του Συμβουλίου. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία ε, ε, θετική για όλους. Πρέπει να προχωρήσει το θέμα αυτό, πρέπει να στηριχθούμε στο χρονοδιάγραμμα που προτείνει ο εισηγητής και νομίζω ότι αν ο πρώτος τριμερής διάλογος εξαγγέλει εν πολύ στο τι θα ακολουθήσει, έχω την αίσθηση ότι θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με επιτυχία. Άλλα σχόλια. Κλοντ, θέλεις να απαντήσεις. Ναι, θα απαντήσω στην κυρία Δοτσέβα ότι για το θέμα της ένταξης, της ενσωμάτωσης, όντως είναι ένα ζωτικό θέμα τα γλωσσικά μαθήματα και έχει υποβάλει μια τροπολογία η συνάδελφος. Δεν υπάρχει στο σώμα ε, εκεί που λέει, αλλά υπάρχει στην έκθεση. Θέλουμε όταν πάμε στην Ολομέλεια φυσικά και να συμπεριλαμβάνουμε και το θέμα της ε, ένταξης. Θα κοιτάξουμε αύριο στη συνεδρίαση που θα έχουμε ισκιώδης να το συμπεριλάβουμε επαρκώς, ώστε να καλυφθεί η συνάδελφος. Ευχαριστούμε, Κλοντ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλα σχόλια. Συνεχίζουμε τότε με το σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 5 είναι οι ελάχιστες απαιτήσει για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκών τρίτων χωρών η απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το περιεχόμενο της ε, παρεχόμενης προστασίας. Εδώ θα έχουμε πάλι παρουσίαση. Την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει το σχέδιο έκθεσης. Και η κυρία Λάμπερτ, που είναι η συγγήτριά μας, ετοίμασε μια οδηγία, ένα σχέδιο. Θα μας δώσει λεπτομέρειες για την ε, οργάνωση των εργασιών πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε και το Συμβούλιο. Πρώτα, η κυρία Λάμπερτ, για να μας κάνει τη δικιά της παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα πω ότι είμαι σύντομη, γιατί κάθε φορά που κάποιο λέει ότι θα είναι σύντομο, τελικά μιλάει 10 φορέ παραπάνω από ό,τι αρχικά πιστεύει ότι θα μιλήσει. Θέλω όμω να σα υπενθυμίσω εδώ το εξή. Είχαμε ένα έγγραφο εργασία, είχαμε το σχέδιο εκθεσή μου και τώρα είμαστε στην εξή κατάσταση. Έχει ανοίξει πόρτα για την υποβολή τροπολογιών και η προθεσμία, θα θυμόσαστε, είναι σήμερα στις 6 το απόγευμα η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Οπότε έχω ήδη πάρει αρκετέ τροπολογίε και φαντάζομαι ότι θα φτάσουν και άλλε μέχρι τι 6 σήμερα. Η χτεσινή μας συνάντηση με την Επιτροπή ήταν πολύ χρήσιμη. γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να τους ρωτήσουμε διάφορες λεπτομέρειες όσον αφορά το περιεχόμενο, όσον αφορά τις επιπτώσεις των προτάσεών μας και των προτάσεων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπενθυμίζω επίση τους Ευρωβουλευτές ότι προβλέπεται σήμερα το μεσημέρι συνεδρίαση με τους συντάκτες του Odysseus Network σχετικά με την μελέτη που έχουν ε, κάνει οι ίδιοι και μας την είχαν υποβάλει κάποια στιγμή εδώ στην Επιτροπή μας, μας τις είχαν παρουσιάσει. Θα γίνει το μεσημέρι. 5ε2 είναι η αίθουσα. Δεν μας δόθηκε ευκαιρία μετά τις 15... μας δόθηκε ευκαιρία να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Θα ήθελα όμως να ακούσω το Συμβούλιο τι προβλέπει όσον αφορά το δικό τους χρονοδιάγραμμα. Γιατί καθυστέρησαν. Νομίζω ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο για αυτή την υπόθεση όπως και για άλλες. Είναι λογικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσει η θέση του να συζητηθεί στο Συμβούλιο και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία, της ημερομηνίας κλπ. Για το περιεχόμενο γίνονται οι συζητήσεις, τα έχουμε ήδη πει, δεν χρειάζεται τώρα να συζητήσουμε πάλι επί της ουσίας. Όμως θέλω το Συμβούλιο τώρα να μιλήσει και να μας πει πώς κινούνται εκείνοι για το θέμα του ασύλου, για παράδειγμα, όπως και για τα άλλα. Ευχαριστούμε κυρία Λάμπερτ. Επιτροπή και Βέλγικη Προεδρία. Ποιος θα πάρει το λόγο. Η κυρία Γκάνγκ, όχι. Η Βελγική Προεδρία. Α, ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Λάμπερτ για την έκθεση την οποία έχουμε πάρει και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια καλή βάση προς Περιμένουμε και τις ε, τελευταίες τροπολογίες. Και την προηγούμενη φορά σχολίασα την ε, έκθεση αυτή, αλλά τώρα με ρωτάτε πώς έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Προχωράνε οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Την προηγούμενη εβδομάδα καταφέραμε να έχουμε τεχνικές συζητήσεις για την υπόθεση αυτή και να ολοκληρωθούν αυτές την ομάδα εργασίας για το άσυλο. Είναι η τελευταία ομάδα εργασίας ουσιαστικά Οπότε, όντω, συζητήσαμε τα τεχνικά ζητήματα και τα ολοκληρώσαμε. Επίση, την προηγούμενη εβδομάδα, σε επίπεδο ε, Επιτροπή ε, Στρατηγική για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επίση συζητήσαμε για το θέμα αυτό. Και παραμένουν ανοιχτά τα εξή θέματα. Πρώτον, ο ορισμός ποια είναι μέλη της οικογένειας και δεύτερον, η προσέγγιση όσον αφορά την προστασία. πρόκειται για δύο περιπτώσεις και θέλουμε να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Αυτή είναι η συζήτηση λοιπόν που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο σε επίπεδο κορεπέρ αυτό το μήνα ή τον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, να συνεχίσουμε και τέλη Νοεμβρίου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε διάλογο με την κυρία Λάμπερτ. Λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση πραγμάτων στο Συμβούλιο. Θέλει κάποιος Ευρωβουλευτής το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Ρομέρο. Κυρία Ρομέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή τροποποίησης είναι ένα κείμενο που έχει ξαναδουλευτεί. Εμείς συμφωνούμε με τη θέση της εισηγήτριας της κυρίας Λαμπέρτ γιατί έχει ήδη συμπεριλάβει τις προτάσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων και σε θα στηρίξουμε τις δικές της τροπολογίες. Δεν υπάρχει χρόνος έτσι κι αλλιώς για να υποβάλουμε νέες τροπολογίες ή να αλλάξουμε τις ήδη υπάρχουσες. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις νομικές παραδόσεις, που βάσει αυτών μερικές φορές τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των γυναικών, εδώ θα έπρεπε να διευκρινίσουμε περισσότερο το θέμα στη νέα εκδοχή της έκθεσης. Είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το κείμενο που μπορεί να τροποποιήσει το Κοινοβούλιο να είναι τόσο μικρό. Είμαστε σε συναπόφαση. Θα έπρεπε να μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλα πιο σημαντικά θέματα. Πάντω μέσα σε αυτό το περιορισμένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορεί να δουλέψει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά να υποβάλουμε πρόταση που να λέει ότι ό,τι νομικές παραδόσεις ή ηθικέθημα που ισχύουν και που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών να ε, εξετάζονται κάθε φορά και να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά που υπάρχει μια αίτηση για άσυλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ρομέρο, λέει ο Πρόεδρος Χολμάγερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τις βασικές μου τοποθετήσεις ως προς την υπόθεση αυτή τις εξέφρασα και στην πρώτη τελευταία συνεδρίαση διεξοδικά, γι' αυτό δεν θα τις επαναλάβω. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λαμπέρτ για την πολύ καλή συνεργασία και για τη διάθεση συνεργασίας. Μία ερώτηση μόνο προς το Συμβούλιο ουσιαστικά μπορεί το Συμβούλιο να μας εξηγήσει ακριβώς πώς ε, έχει η κατάσταση σχετική με την επανένωση με τα μέλη της οικογένειας και αν υπάρχει επαρκής ε, προστασία, ποια είναι η κατάσταση στη συζητήση του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κυρία Κιγιώμα. Δύο λόγια μόνο. Η κυρία Λαμπέρ μπορεί να λέει ότι θα μιλήσει σύντομα, αλλά είπε αρκετά νομίζω. Ε, λέμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση της Επιτροπής. Θα πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις της τρέχουσας ε, νομοθεσίας. Και μια και το ανέφερε και ο κύριος από το Συμβούλιο, ως προς τη σημασία των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους παραδοσιακούς πρόσφυγες και σε εκείνους στους οποίους προσφέρεται η επικουρική ε, βοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να επιμείνω ιδιαίτερος, διότι είναι απαραίτητο να μην επιτραπεί στα κράτη-μέλη να αρνούνται την συμπληρωματική, την επικουρική αυτή ε, προστασία πέραν της συμβατικής, των προσφέρουν συνθήκες δηλαδή. Και έτσι θα μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε ίσω και το κόστος ορισμένων διαδικασιών. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Λάμπερτ για τη δουλειά τη και την ενημερώνω ότι σκοπεύω να καταθέσω δύο τροπολογίες, μία για το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και μία για την έννοια του παράγοντα προστασία. Ω προ το πεδίο εφαρμογή θεωρώ ότι πρέπει να διευρυνθεί για να καλύπτει όχι μόνο τους υπηκόους τρίτων κρατών που θα, υποθέσουν, θα καταθέσουν μια αίτηση για χορήγηση ασύλου, γιατί η συνθήκη της Γενέβης δεν ορίζει ή δεν επιτρέπει καλύτερα περιορισμό για λόγους γεωγραφικούς ή καταγωγής. Εν πάση περιπτώσει όμω αυτό επί τη ουσία μπορούμε να το συζητήσουμε. Και δεύτερο για τον παράγοντα ή το φορέα προστασία που θα πρέπει αποκλειστικά να είναι οι εθνικές αρχές, κατά την άποψή μου. Διότι κόμματα οι οργανώσεις, με όση βέβαια αξία και να έχει δουλειά τους, δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν το σεβασμό του κράτους δικαίου και να προσφέρουν αποτελεσματική και διαρκή μακροπρόθεσμα προστασία. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ξανασυστήσουμε με την κυρία Συγγετρία. Ευχαριστώ κύριε Μπρόνς. Πρόεδρε, ε, σήμερα το πρωί ακούμε πράγματα που έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Αυτό που θα δικαιούται το άσυλο θα πρέπει να είναι όχι μόνο αυτό ο οποίο κινδυνεύει προσωπικά, που βρίσκεται εκτεθειμένος δηλαδή, αλλά ή οσδήποτε κινδυνεύει να αποσταλεί σε μια χώρα επικίνδυνη, δηλαδή βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της επικινδυνότητας της χώρας. Εάν δεχθούμε λοιπόν αυτό ως βασική αρχή θα πρέπει να καταλήξουμε και στη λογική της ε, συνέπεια ότι εφόσον είναι απαράδεκτο το να ε, αποστέλουμε σε χώρες επικίνδυνες εκείνους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερες περιπτώσεις, τότε θα πρέπει να δεχθούμε ε, την παραμονή όλων αυτών των πολιτών των επικίνδυνων χωρών εντός των σύνορων τους. Δηλαδή θα πρέπει να φέρουμε όλους τους Κινέζους, όλους τους Πακιστανούς και δεν ξέρω ποιους άλλους. Νομίζω ότι είναι αρκετά για σήμερα το πρωί, Πρόεδρε. Αρκετά ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ε, κυρία Λαμπέρτ, ακούσαμε και από, την Προεδρία και από τους βουλευτές. Θέλετε να επανέλθετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η αρχή της μη ε, αναπομπής είναι βασική αρχή του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι ζήτημα κοινοβουλίου φυσικά να την ανατρέψει. Επίσης, συζητήσαμε τους περιορισμούς ως προς την ε, επαναδιατύπωση της ε, οδηγίας. Ακούσαμε τις θέσεις του Συμβουλίου σε σχέση με τις προτάσεις ε, συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο εύκολο και στι διαπραγματεύσει. Εν πάση περιπτώσει, με χαρά θα δω τι τροπολογίε σα. Πέραν αυτών τις οποίες έχω ήδη λάβει. Ε, Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε με τους κοιόδη ηγητέ και βέβαια και στην Επιτροπή μα 15 του μηνός. Ευχαριστώ. Thank you. And as... Ευχαριστώ πολύ. Για δε το ερώτημα της κυρίας Χόλμαϊερ. Θα έχει την καλοσύνη να απαντήσει η Προεδρία. Ευχαριστώ. Με ρωτήσατε για τον ορισμό τι είναι μέλος της οικογένειας. Όπως σας είπα, είναι κάτι που συζητιέται στο Συμβούλιο. Δεν μπορώ εγώ να προκαταλάβω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Αρχικά, η Επιτροπή του Συμβουλίου συζήτησε, συνέχισε τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα όπως σας είπα, αλλά δεν μπορώ να προκαταλάβω πού θα καταλήξει αυτό το θέμα για το τι είναι μέλος της οικογένειας. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι το σημείο 6. που είναι η εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα και τη θέσπιση άδεια εξαγωγή καθώ και το μέτρο εισαγωγή και διαμετακόμιση για πυροβόλα όπλα, μέρη του και εξαρτήματά του, όπω επίση και πυρομαχικά. Είμαστε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σε παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης αυτής είναι η συνάδελφός μας, η κυρία Ματιέ. Έχουμε πρόταση της Επιτροπής που μιλάει για την εφαρμογή του άρθρου 10 των ε, Ηνωμένων Εθνών, του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη ε, επί της ουσίας. Ζητήθηκε από τη Λίμπα να συνεργαστεί βάσει το άρθρο 50 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Μαρίνη πρώτα απ' όλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει την πρόταση αυτή, μετά στη Βέλγικη Προεδρία για να μας παρουσιάσει την κατάσταση πραγμάτων στο Συμβούλιο. Και μετά θα ξεκινήσουμε συζήτηση. Κύριε Μαρίνη. Διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε το πρωτόκολλο αυτό για τα πυροβόλα όπλα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα προσαρτημένο διεθνές έγγραφο στα πλαίσια της νομικής τάξης των Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα πρέπει να μεταφέρει τις προβλέψεις αυτές στην κοινοτική νομοθεσία. Τα άρθρα τα οποία αφορούν την εσωτερική αγορά αντιμετωπίστηκαν το 2008 με την οδηγία για την εσωτερική αγορά. Το άρθρο 10 προβλέπει τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εμπορική πολιτική και εκεί τα κράτη-μέλη δεν έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. δεν έχει επικυρωθεί η διεθνής αυτή συμφωνία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμως μια διεθνής υποχρέωση την οποία έχει αναλάβει για την παρεμπόδιση της διάδοσης των μικρών πυροβόλων όπλων στον κόσμο. Τα άρθρα 207 και 346 της συνθήκης προβλέπουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο στα πλαίσια του οποίου ακριβώς θα εφαρμοστεί το νέο άρθρο 10. Η πρόταση καταρχάς θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει του συγκεκριμένου άρθρου και επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσει του άρθρου 346 που αναφέρεται στα θέματα εθνικής ασφαλείας των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να, αναλαμβάνει, να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλειά του και γι' αυτό ακριβώς η πρόταση αυτή ε, ε, δεν είναι κάτι το οποίο καλύπτει τις στρατιωτικές χρήσεις των όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να φέρει πέρα στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η εναρμόνιση που απαιτείται στα πλαίσια της κοινή εμπορικής πολιτικής, στα πλαίσια της εξαγωγής πυροβόλων όπλων για πολιτική χρήση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή των μέτρων τα οποία μπορεί να λάβει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει επίσης και τις προτάσεις του πρωτοκόλου ε, για το, ε, για, την, ε, για τα μικρά όπλα. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης προτείνει την διαδικασία να συνεχιστεί στα πλαίσια των πρωτοβουλειών των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια ε, μεγάλη προπαρασκευαστική μελέτη η μελέτη επιπτώσεων έχει βασιστεί στις διαπιστώσεις του 2006 και 7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλους τους εμπλεκομένους που εκπροσωπούν τις διάφορες ομάδες συμφερόντων όπως την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών Όπλων, το εμπόριο για πολιτική χρήση όπλων και τα κτλ. Έγιναν δύο συναντήσει συναντήσεις στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2007 στις οποίες πήραν μέρος και μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ανοίξαμε και ένα λογαριασμό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για μια συνέχιση της διαβούλευσης. Η διαβούλευση λοιπόν απευθύνεται κυρίως ε, στα κράτη-μέλη και 19 από τις 27 χώρες έστειλαν απαντήσεις και πήραν μέρος στις συναντήσεις και ενεπλάκησαν με τον ένα τρόπο ή τον άλλον. Σχετικά με την διαβούλευση ιδιωτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε μια αρκετά μεγάλη διαβούλευση. Αποστήλαμε ερωτηματολόγια ε, Εμπλεκομένου στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γνώμες οι οποίες εκφράστηκαν στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής περιλαμβάνονται ε, στο έγγραφο το τελικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν ο κανονισμός δεν γίνει δεκτός, η κατάσταση ε, θα παραμείνει στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δεν θα καλυφθούν και οι προβλέψεις του πρωτοκόλου των Ηνωμένων Εθνών δεν θα εφαρμοστούν. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να τιμήσει θα λέγαμε τις ανηλυμένες της υποχρεώσεις προς τη διεθνή κοινότητα. Όπως σας είπα προηγουμένως, η πρόταση λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για απλουστευμένα μέτρα για προσωρινές αδειοδοτήσεις εξαγωγών, για τη μετρίαση των αρνητικών επιπτώσεων των μέτρων εφαρμογής του πρωτοκόλου για μικρά όπλα, την χρήση πολλαπλών αδειοδοτήσεων για πολλαπλές αποστολές προϊόντων, όπως επίσης και προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την έκδοση της άδειας εξαγωγής. Νομίζω ότι έχουμε κάνει σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση αρκετά ισορροπημένη που καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων. Δεν θέλησαμε να δημιουργήσουμε νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προς στιγμή δεν έχω να πω, προς στιγμή, συγγνώμη, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι. Είμαι όμως στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, κύριε Μαρίνα. Ας ακούσουμε τώρα τη Βελική Προεδρία. Θέλει το λόγο η Προεδρία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στόχος της Προεδρίας είναι να ολοκληρωθεί η τεχνική επεξεργασία του θέματος πριν τη λήξη της Προεδρίας μας. Εξετάζουμε άρθρο προς άρθρο την πρόταση και θα συνεχίσουμε στις τέσσερις υπόλοιπες συνεδριάσεις που έχουμε στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you. Now, let's hear... Καλώς. Ας ακούσουμε τους ευρωβουλευτές τώρα. Έχουμε την συγκεντρία, την κυρία Ματιέ. Παρακαλώ κυρία Ματιέ. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και να εξασφαλίσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες σιγουριά και ασφάλεια, η Επιτροπή προτείνει την ε, επικύρωση του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα και προτείνει έναν κανονισμό με συναπόφαση και το Κοινοβούλιο θα μάλλον έχει επιλέξει το άρθρο 5 για να βάλει τις δύο επιτροπές ΣΥΝΤΑ και ΛΥΜΠΕ να συνεργαστούν. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για όπλα, ελαφρά όπλα, ε, που δεν περιλαμβάνουν τα στρατιωτικά όπλα ή τα όπλα της αστυνομίας. Απευθύνεται λοιπόν στους ε, κοινούς χρήστες που μπορεί να είναι κυνηγοί αλλά μπορεί να είναι άλλοι οι οποίοι ως άθλημα έχουν ε, τη σκοποβολή, γιατί ξέρουμε ότι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε τέτοιου είδους αθλήματα. Οι αθλητές αυτοί είναι πάρα πολύ συμπαθητικοί και γι' αυτό λοιπόν κάνει μια πολύ καλή πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει να κάνει με την απλοποιημένη διαδικασία άρθρο 7.5 και επίσης η πρόταση αυτή έχει να κάνει και με την έκθεση, την πραγματογνωμοσύνη και την ε, επισκευή πυροβόλων όπλων. Βέβαια θέλω ο κύριος Μαρίνη να μου το επιβεβαιώσει αυτό, γιατί διαβάζοντας την πρόταση της Επιτροπής για αυτά τα τρία σημεία, δηλαδή την πραγματογνωμοσύνη, την έκθεση και την επισκευή, τα πράγματα μου φαίνονται όχι πολύ συγκεκριμένα, λίγο φλού κύριε Μαρίνη. Στην πρόταση αυτή κανονισμού είπαμε ότι έχει να κάνει με τους αθλητές στη σκοποβολή, με τους κυνηγού. Ε, για αυτούς πρέπει να κατασκευάζονται όπλα και να πολλούνται. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν μόνο μεγάλες μονάδες παραγωγής τέτοιων όπλων, υπάρχουν και μικρά τελειέ. Και υπάρχουν και εξαγωγές βέβαια μετά των όπλων προς τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν από αυτού έκανε μια μελέτη αντικτύπου για την πρόταση αυτή. Και εδώ ανησυχώ κύριε Μαρίνη, γιατί το εύρος στο οποίο βασίζεται η πρότασή σας είναι 1350 ευρώ, ενώ στην άλλη περίπτωση είναι 1.600. Πρέπει να ξέρουμε ότι κανείς εδώ δεν αμφισβητεί ότι στόχος μας είναι η ασφάλεια αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κόστος εδώ και θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα γιατί σήμερα που είμαστε σε περίοδο κρίσης και προσπαθούμε να εκπονήσουμε τη στρατηγική μας για το 2020 καταλαβαίνετε ότι πολύ θα ήθελα να βρούμε ένα μεσόρο. Δηλαδή αυτοί που κατασκευάζουν ή που εξάγουν τα όπλα να μην επομίζονται από μόνοι τους το κόστος της ασφάλειας το οποίο εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει. Η συνεργασία μου με τους κοιόδες εισηγητές ήταν πάρα πολύ καλή. Περιμένω τώρα τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Άκουσα την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Μαρίνη Έχω ήδη συναντηθεί μαζί του, μιας και είμαι υπεύθυνο για την έκθεση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε στην Επιτροπή Ίντε. Είχαμε συναντήσεις και με το Συμβούλιο και μου φαίνεται ότι το έγγραφο είναι αρκετά ισόρροπο και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από τα διάφορα όργανα Φυσικά και περαιτέρω ε, βελτιώσεις είναι πιθανές. Ε, μπορώ να σταθώ σε δύο θέματα τώρα. Το πρώτο είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών των σχετικών με τα καθεστώτα δανειοδότησης. Και από την άλλη, αυτή στιγμή ε, γίνει δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση, το παρόν σύστημα το οποίο ε, χαρακτηρίζεται από χώρες που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει, χώρες που έχουν υπογράψει και επικυρώσει και χώρες που δεν έχουν κάνει τίποτα από τα δύο. Υπάρχει μια σύγχυση ενώ όταν προχωρήσουμε στην έκθεση αυτή θα έχουμε ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για το σύνολο της Ένωσης. Το είπε αυτό η κυρία Ματιέ αφορά τα μικρά πυροβόλα όπλα, αφορά όμως επίσης και μία μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία τέτοιων όπλων διαφορετική από τα πολεμικά. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με ό,τι έχει σχέση τα πολεμικά όπλα, αλλά μιλάμε για αγωνιστικά όπλα, όπλα σκοποβολής και κυνηγίου. Ένας τομέας ο οποίος ε, εκπροσωπεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα σημαντικά, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ. Έχω μια κάπως διαφορετική προσέγγιση. Γιατί δεν ε, αντιλαμβάνομαι ακριβώς ε, τον αναψυκτικό χαρακτήρα, τον ε, διασκεδαστικό χαρακτήρα της χρήσης των όπλων. σας μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Επίσης, γιατί δεν βλέπω δύο, γιατί υπάρχουν διαφορετικές επιλογές από την μελέτη επιπτώσεων και επίσης διότι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να επικρατήσουν οι στόχοι του άρθρου 10 της Συμφωνίας των Αθηνών. Ε, έστω και αν λέμε ότι θέλουμε ψυχαγωγική χρήση ή αθλητική χρήση των όπλων, γιατί να κυκλοφορούν όπλα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω επίσης είναι γιατί έρχεται με τόση καθυστέρηση αυτή η πρόταση, όταν έχουμε ήδη από το 2002 αυτή την ε, ε, πρώτη ιδέα τέλο πάντων, το 2005 μόνο η η πρόταση οδηγίας, φαίνεται ότι θα μπορούν ε, οι κυνηγοί με μία άδεια που ισχύει σε μία χώρα να πηγαίνουν σε άλλη χώρα στις οποίες δεν έχουν άδεια. Το οποίο σημαίνει ουσιαστικά δικαίωμα οπλοχρησίας, οπλοκατοχής και οπλοχρησίας ε, χωρίς άδεια. Θα ήθελα να ενημερωθώ επίση για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει με τι οποίε έχετε διαβουλευθεί, διότι έχω την εντύπωση ότι είναι κάπω μονομερεί οι απόψει που εκφράζουν. Και εάν ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο 10 της προτάσεως, τους ε, κυνηγούς και σκοπευτές για αθλητικούς ε, λόγους ε, λέτε ότι θα τους καταγράφετε για ένα ορισμένο διάστημα κλπ. Για πόσο καιρό θα μένουν τα στοιχεία αυτά καταχωρημένα. Αυτά ε, ζητώ συγγνώμη που θα χρειαστεί να φύγω πριν να ακούσω τις απαντήσεις σας, αλλά παρακαλώ δώστε τις απαντήσεις γιατί θα ενημερωθώ εγώ όπως πρέπει. Ο κύριος Λιτσιού. Ευχαριστώ. Το πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται στα μη στρατιωτικά όπλα. Μη πολεμικά όπλα. Έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί χρησιμοποιείται ένα μόνο άρθρο σαν ε, νομική βάση. Και το λέω αυτό κυρίω γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με την κοινή εμπορική πολιτική και το άρθρο 10 του Πρωτοκόλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβολόπλα έχει να κάνει με την πρόληψη του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να είχαμε βρει μια άλλη νομική βάση και όχι μόνο αυτό το άρθρο. Γνωρίζω πολύ καλά τον τομέα. Και μπορώ να σας πω ότι σε κάθε κράτος μέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης, υπάρχουν ε, πολύ αυστηροί κανόνες όσον αφορά την παραγωγή, την εμπορία και την κατοχή πυροβόλων όπλων. Κάθε κράτος μέλος έχει πολύ αυστηρά μέτρα. Ο κανονισμός αυτός λοιπόν δεν λαμβάνει υπόψη την επικουρικότητα. Υπογραμμίζει μόνο την πτυχή κοινή πολιτική. Γι' αυτό αναρωτιέμαι, γιατί να μην έχουμε μια οδηγία καλύτερα για να μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και τι ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια από συνάδελφο. Θέλει κανείς άλλος συνάδελφος να σχολιάσει. Ας απαντήσει ο κύριος Μαρίνη, παρακαλώ, από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ με τις παρατηρήσεις κυρίας Ματιού ως προς τις ε, συνέπειες του καλωσμού αυτού με την αποστευμένη διαδικασία. Όπως είπα και στις αρχές μου παρατηρήσεις, προσπαθούμε να εισαγάγουμε απλουστευμένες διαδικασίες, έτσι ώστε να μην ε, επιβαρυνθεί πολύ η διαδικασία θα αντιμετωπίσουν όσοι νόμιμα χρησιμοποιούν τα όπλα. Οι επιστευμένε λοιπόν διαδικασίε του άρθρου 7 προβλέπονται για κάθε περίπτωση, για τον κυνηγό, για τον σκοπευτή, για τον αθλητή σκοποβολής, στην διαμετακόμιση κτλ. Για όλους λοιπόν. Από την άλλη και για τους λόγους που έχουν, και για λόγους που έχουν επισημάνει τα Υπουργεία των Εσωτερικών διαφορών κρατών μελών, για τις εξαγωγές απλουστεύουμε τη δικασία μόνο για τους αθλητικούς σκοπευτές και τους κυνηγού, αλλά όχι για την ε, ε, επισκευή και έκδοση. Αυτά για λόγους ασφάλειας. Όσον αφορά το κόστος του, ε, της μελέτης αξιολόγησης των επιπτώσεων, εκτιμούμε ότι αντιστοιχεί στο 0,19% της όλης αξίας εξαγωγών όπλων, πυροβόλων όπλων για το 2009. Αυτό θα ήταν, το, η επιπλέον επιβάρυνση που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία. Τη βρίσκουμε πολύ μικρή. Και αυτά χάρη σε μία μέθοδο υπολογισμού που εκπονήσαμε και πρέπει να σας πω δεν ήταν καθόλου εύκολο να την εξασφαλίσουμε αυτή τη μέθοδο. Όσον αφορά το λόγο για τον οποίο ήρθαμε τώρα μόλις να αναφερθούμε στον κανονισμό αυτό και γιατί η Επιτροπή υποβάλλει τον κανονισμό αυτό μόλις σήμερα. Ήθελα να εξηγήσω ότι χρειάστηκε να αναμένουμε την έγκριση της οδηγίας που δημιουργούσε το αντίστοιχο τμήμα της εσωτερικής αγοράς. Και μετά μόνο μπορούσε το πρωτόκολλο 10 να υποβληθεί στη διαδικασία αυτή από την Επιτροπή. Χρειάστηκε να περάσει όλη η διαδικασία της μεταφοράς του Εθνικού δίκαιο των διαφόρων κανόνων που προέβλεπε το πρωτόκολλο στην κοινοτική νομοθεσία. Με πρώτο στάδιο την ε, διαπραγμάτευση και έγκριση της οδηγίας κατά το 2008 που καλύπτει το τμήμα που αντιστοιχεί στην εσωτερική αγορά. Και μετά ασχοληθήκαμε με το μόνο άρθρο το οποίο έμενε εκτός αυτής της οδηγίας, το άρθρο 10. Ο κανονισμός δηλαδή στηρίζεται και αυτός σε μέτρα και αρχές που ήδη ακολουθεί η οδηγία του 2008. Όπως σε παραδείγματα, τους ορισμούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί βέβαια η συνοχή των όσων έχουμε προσδιορίσει νομοθετικά σε εσωτερικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ε, των όσων προσδιορίζουμε στις εξωτερικές μας σχέσεις με τρίτες χώρες. Η νομική βάση είναι το παλαιό άρθρο 133. Το τωρινό 207, εξωτερικό εμπόριο. Αυτή είναι η εξωτερική, ε, η νομική βάση, η οποία είχε προσδιοριστεί από την αρχική εντολή διαπραγμάτευσης που είχε χορηγήσει το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης του πρωτοκόλλου. Βάσει λοιπόν αυτής της νομικής βάσης και σε σχέση συγκεκριμένα με το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου η Επιτροπή υποχρεούται να ακολουθήσει ως νομοθέτημα τη λύση του κανονισμού, γιατί αυτό επιβάλλει το άρθρο 207. Ως προς την μελέτη των επιπτώσεων, που έλεγα και στην πρώτη παρέμβαση, υπήρξε μια, μια μακρά σειρά διαβουλεύσεων με διαφόρους παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο και έχουμε ιδιαίτερως ε, συμπεριλάβει στην μελέτη ε, ε, επιπτώσεων τον κατάλογο όλων των εμπλεκομένων και οργανώσεων που συμμετέσχουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Επίσης και μια τελευταία παρατήρηση. Εδώ δεν προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα προσώπων με το νομοθέτημα αυτό. Με το νομοθέτημα αυτό. Απλώς εξυπηρετούμε το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκει το νομοθέτημα. Δηλαδή το δικαίωμα της το δυνατότητα χνηλασίας αυτών των πυροβόλων. Δυνατότητα χνηλασίας την οποία θεωρούμε ε, θεμελιώδους σημασίας έτσι ώστε να μην αφαιθεί ελεύθερο το πεδίο για παράνομη διακίνηση όπλων, δηλαδή για να μην χρησιμοποιούνται για λόγους παράνομους, για σκοπούς παράνομους τα όπλα αυτά. Αυτή ήταν η πηγή έμπνευση για αυτόν τον κανονισμό, όπως και, όλων των πρωτοκόλων, όπως και για όλα τα πρωτόκολλα των ΗΕ. Και προσπαθούμε την αρχή αυτή να την μεταθέσουμε, να τη μεταφέρουμε στην κοινοτική νομοθεσία, διαφυλάσσοντας και ως βασική αρχή, ως βασικό μέλημα, την ανάγκη να μην επιβαρυνθούν υπερβολικά οι διαδικασίες. Δηλαδή τελικά ο χρήστης και ο εξαγωγέας όπλων. Όποιος το πράττει βέβαια για λόγους, για σκοπούς νόμιμους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Thank you for the explanations. If Άλλα σχόλια. Η κυρία Ματιέ, μήπω, η συγγήτρια. Όχι. Τότε. Να σταματήσουμε για πέντε λεπτά. Γιατί τώρα κυκλοφορεί ο κατάλογος ψηφοφοριών με τις τελευταίες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί επί της ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε την πρωτοβουλία πολιτών. Ο κατάλογος ψηφοφορίας κυκλοφορεί, οπότε πέντε λεπτά χρειάζονται ακόμα μέχρι να έχετε όλοι στα χέρια σας τον κατάλογο αυτόν. Θα ξεκινήσουμε σε 5 λεπτά ακριβώς την ψηφοφορία. Dear colleagues, if you're all set, we may get started. Okay. Λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Έχουμε μια μεγάλη ψηφοφορία. Θα μας πάρει δηλαδή χρόνο. Έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες. Πρώτα, η πιο σημαντική ψηφοφορία για σήμερα το πρωί είναι εκείνη που αφορά την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Οι συγγήτριε είναι οι συνάδελφοι Κίνκα Γκόνς και Σεσίλια Βίλκστρομ. Λοιπόν, εφόσον έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας, την τελευταία εκδοχή, με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις, εφόσον όλοι έχετε αυτό τον κατάλογο, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 70 κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. I mean, that is precisely why we need... Να, γι' αυτό και πρέπει να έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο κατάλογο ψηφοφορίας για να ξέρουμε αν πρέπει να ψηφίσουμε εδώ ή όχι. Λοιπόν, τροπολογία 70. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το τμήμα 3 καταπίπτει και ερχόμαστε στο τμήμα 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 71. Ψηφίστε παρακαλώ. Να αρχίσει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί. Μήπω να αλλάξετε θέση. Αλλιώς θα μετρήσουμε μία ψήφο υπέρ επιπλέον. 25 υπέρ, 23 κατά είναι το αποτέλεσμα. Εσείς τι, κατά ψηφίσατε. Υπέρ, υπέρ, ωραία. Άρα έχουμε δύο ψήφους υπέρ επιπλέον. Οπότε είναι 27 τα υπέρ, 23 οι ψήφοι κατά. Οπότε γκρίνεται. 73. Όχι, 74 διορθώνω ο πρόεδρος. Τροπολογία 74, 75 και 76 για την ίδιες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογίες 12 και 77 μαζί υπέρ. Κατά αποχές Να ελέγξουμε καλύτερα, λέει ο πρόεδρος. 12 και 77 που είναι τις ψηφίζουμε μαζί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Άλντε. Έχει ψηφίσει ένας παραπάνω.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 29 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Εγκρίνονται. 78 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Με προφορική τροποποίηση. 79 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. 80 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 και 83 που είναι ίδιες μαζί λοιπόν. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτονται. Η 14 αποσύρθηκε. 84 υπέρ, καταπίπτει. Οι 82 και 83 εγκρίθηκαν. Όχι, απορρίφθηκαν. Οπότε ψηφίζουμε την 84 τώρα. Υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Κατά τμήματα ψηφοφορία εδώ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. Να ελέγξουμε, εντάξει, θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 87. Ξεκινάει η ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 24 κατά εγκρίνεται. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Θέλατε να έχετε ψηφίσει ναι, οπότε εγκρίνεται. 88 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 89, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 με προφορική τροποποίηση του κ. Ντεγιόγκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε για τη συμβαστική τροπολογία 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 29 ψήφοι υπέρ, 17 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. 17 τώρα, τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω. Αλλά σε ελέγξουμε. 17 λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Much of a stress going on here? Eh? Yes? We're repeating. Να επαναλάβουμε. Δούλεψε, εντάξει. Α. Οπότε, αποτέλεσμα. 24 ψήφοι υπέρ, 22 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται η δεκατά. Τώρα, 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 93. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. ψηφοφορία. 25 υπέρ, 21 ψήφι κατά, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία για την τροπολογία 94. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 18. Ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά λοιπόν ελέγχουμε για την 95. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 24-24. Απορρίπτεται συνεπώς. Αυτό σημαίνει ισοψηφία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε και πάλι. 19. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 96 τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 20. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 με προφορική τροποποίηση. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100. Με προφορική τροποποίηση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 100. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 και 105 τώρα που είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107. Α, όχι, καταπίπτει, διορθώνει ο πρόεδρος. Και φτάνουμε στην 110. Ψηφίσουμε την τροπολογία 110. Σωστά. Ίσως εγώ να έχω λάθος κατάλογο, αλλά για μένα μόνο 106 καταπίπτει. Δεν βλέπω να καταπίπτουν κι άλλες, 107, 108 κλπ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, εγώ δεν το έχω δει καλά. Λέει η κυρία Σκνετίνη. Εντάξει, η 110 έχει τώρα σειρά. Ψηφίζουμε την 110. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, επόμενε καταπίπτουν, 23, 111, 24, 25, φτάνουμε στην 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επόμενες καταπίπτουν και έτσι φτάνουμε στην τροπολογία 117. Με προφορική τροποποίηση. 117 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε. 121. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. 122 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Η Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 123. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 25-25 είναι το αποτέλεσμα, απορρίπτεται συνεπώς. 124 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 τώρα, με κατατμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα της 126 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 27. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της προφορίες. 25 υπέρ. 19 κατά. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι θα ελέγξουμε. 127 λοιπόν. Ψηφίστε. Πέρα στις προφορίες. 27 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 και 132 είναι ίδιες. Τις ψηφίσουμε μαζί, λοιπόν, 28 και 132 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για αυτές τις δύο. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 31 ψήφι υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε μαζί την 134 και την 135 και την ίδια. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 136 με προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και έτσι πάμε στην τροπολογία 30. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 30 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 30. Τροπολογία 30 ψηφίζουμε. Ελέγχουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 28 ψήφι υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 141 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 142 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 τώρα, με κατατμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 32. Ψηφίστε παρακαλώ. τη 24 ψήφοι 23 κατά. Εγκρίνεται. 33 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και έτσι καταπίπτουν οι επόμενες και φτάνουμε στην τροπολογία 2 και 37 που είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις τροπολογίες 2 και 37 που είναι ίδιες. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 38 με προφορική τροποποίηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 με κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται, έτσι δεν είναι, ναι. Τροπολογία. Να ελέγξουμε. Καλά. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 39. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Ναι, απορρίπτεται. 19 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία, η 3 έχει αποσυρθεί. 40. Με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι επόμενες καταπίπτουν. 43 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, θα ελέγξουμε για τη 43. Ψηφίστε παρακαλώ, 43. Πέρας της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω, αλλά αν κάποιο θέλει να ελέγξουν... Όχι. Λοιπόν, 44. Ναι. Πρέπει να την ψηφίσουμε, γιατί απορρίφθηκε 4. 44 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Τροπολογία 44. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της 28 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική... Α, όχι. Διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την τροπολογία 5 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά ας ελέγξουμε. 11. Λοιπόν, ηλεκτρονικά παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 19 κατά εγκρίνεται. Τώρα, φτάνουμε στη 49 έτσι. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα τη 49. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. 28 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 50 και την 51 μαζί για την ίδια. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι 7 και 52 καταπίπτουν. 53 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτεται. Που σημαίνει ότι ψηφίσουμε την 54 τώρα. Υπέρ. κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Τροπολογία 54. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται. 8. Πρέπει να την ψηφίσουμε ακόμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του κύριου Ένσιου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την προφορική τροπολογία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της προφορίας. 27 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε γιατί νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι όπως και με το δεύτερο τμήμα, αλλά σε ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. 25-25. Απορρίπτεται δηλαδή. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 60 έχει αποσυρθεί. 61 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά για την τροπολογία 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τελική ψηφοφορία για το τροποποιημένο πια κείμενο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 48 υπέρ, καμία ψήφος κατά. Συνεπώς εγκρίνεται και συγχαρητήρια στις εισηγήτριες King Gagons και Cecilia Wildstrom. Thank you all. Now we're moving to the following vote because this electronic vote has not come to an end yet. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση έκθεσης Διακόπτει ο Πρόεδρος. Yes. We voting. Please. Dear colleagues. about to finish. Συνάδελφοι, θα τελειώσουμε όπου να είναι, αλλά δεν έχουμε ακόμα τελειώσει ακριβώς. Παρακαλώ καθίστε και συγκεντρώστε την προσοχή σας στην ψηφοφορία proposal for the of σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γεωργία για την επανεισδοχή ε, προσώπων οι οποίοι ε, βρίσκονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τα κατάλληλη άδεια. Γεωργία draft recommendation. We're having an electronic vote. Λοιπόν, η ηλεκτρονική ψήφος ε, για την πρόταση σύστασης, δεν υπάρχουν τροπολογίες, ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας, «42 υπέρ, 6 κατά, γίνεται δεκτή η σύσταση». Μια επεξήγηση ψήφου έχουμε. Θα διαβάσω την επεξήγηση ψήφου. Ναι, αν θέλετε, ναι. Όχι, λένε οι υπόλοιποι. Έτσι και αλλιώς το έχουμε ετοιμάσει γραπτά, το κείμενο θα σας το υποβάλουμε. Καλώς. Θα περάσουμε τώρα στην πρόταση σύστασης για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γεωργία για τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων. Η κυρία Γκρισμπέκ είναι η συγγήτρια. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες, οπότε ψηφίζουμε απευθείας. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. 47 υπέρ, 1 κατά. Για μια ακόμη φορά συγχαίρουμε την κυρία Γκρισμπέκ. Το κείμενο γίνεται δεκτό. Έχουμε τώρα την πρόταση έκθεσης ε, για, τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο των τρίτων χωρών που θα πρέπει οι ε, πολίτες τους να έχουν θεώρηση όταν ε, διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών και ποιοι είναι οι πολίτες οι οποίοι εξαιρούνται αυτής της απέτηση. Ο Διάστε Μέρα είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι στην αιτιολογική σκέψη έχουν γίνει κάποιες τεχνικές τροποποίησεις, μικρές. Εδώ μιλάμε για 130 νομοθέτες, ενώ στο πρώτο τρίμηνο μιλούσαμε για μια ανάπτυξη της Ταϊουάν 13,27%. Θα ήθελα πάντως, Πρόεδρε, εδώ να σας αναφέρω το εξή Το περιεχόμενο της επιστολής της 8 Οκτωβρίου από το Διευθυντή του Γραφείου του Σταϊπέ της Βρυξέλλες, το Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην ε, Προεδρία του Συμβουλίου και στους εκπροσώπους Βουλγαρίας, Κύπρου και Ρουμανίας, όπως και εσείς ο ίδιος ε, έχετε επιστολή και εγώ. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνησή μου αποφάσισε να αφαιρέσει τα σχετικά με τις θεωρήσεις για τη Ρουμανία και την Κύπρο μέχρι 30 μέρες γύρω στην Ταϊωάν μέχρι ε, τον Ιούλιο του 2010. Έτσι λοιπόν σταματάνε οι θεωρήσεις βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας και προσφέρεται σε όλους τους πολίτες ε, του Σέγγεν και στους πολίτες της Κύπρου και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για 90 μέρες παραμονή. Και το ίδιο ισχύει για τον χώρο Σέγγεν όσον αφορά τους πολίτες από την Ταϊβάν. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε, κύριε Διαθεμέρα. Για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης της Ταϊβάν. Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την έκθεση. Πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την τροπολογία του εισηγητή και μετά το τροποποιημένο κείμενο. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία όμως θα ψηφίσουμε. Α, όχι, όχι ηλεκτρονικά την τροπολογία, διορθώνει ο πρόεδρος. Συγγνώμη. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτή τη φορά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Πέρα στις 47 υπέρ, 1 κατά. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια κύριε Δίες Δεμέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας στην ψηφοφορία. Και τώρα, περνώ στο επόμενο θέμα. Το υπαριθμό 11. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. έχει αναβληθεί ήδη μία φορά και έχει να κάνει με την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Frontex δηλαδή. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ θερμά να διατηρήσετε την ησυχία, να συγκεντρωθείτε στη δουλειά. Βλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι αποχωρούν. Σας εκλυπαρώ λοιπόν. Ησυχία. Να συγκεντρωθούμε στο θέμα μας. Σημείο 11. Σας παρακαλώ If you're Παρακαλώ. Έχουμε εδώ προβλέψει μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων στην ημερήσια διάταξη. Σε σχέση με την αναθεώρηση της εντολής της υπηρεσίας Frontex. Ξέρετε ότι η αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών επισκέφθηκε πριν από ένα μήνα τη Frontex και στη συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια στι 4 Οκτωβρίου επίσης συστήθηκε το θέμα αυτό. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Μπουσούτιλ, τον εισηγητή. Για να ακούσουμε την παρουσίασή του, τις νέες εξελίξεις. Μετά θα μας μιλήσει η Βελγική Προεδρία και η Επιτροπή, εφόσον επιθυμώ να λάβουν το λόγο, για να μας ενημερώσουν και εκείνους με την πλευρά τους για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη Frontex. Πρώτα όμως, παρακαλώ, να ακούσουμε τον κύριο Πουσούτη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πολύ σύντομα, οι τελευταίες εξελίξεις. προκειμένου και μια ανταλλαγή απόψεων. Ε, πρώτη, ουσιαστικά δεν είχε καταστεί δυνατή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων, γιατί ε, διαγράφηκε από την ημερήσια διάταξη ε, λόγω ε, πολύ φορτωμένου προγράμματο. Πρώτη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων τώρα και παρακαλώ του συναδέλφου να συμμετάσχουν και να δώσουν τι πληροφορίε του, τι ιδέε του στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Έχουμε μέχρι στιγμή δύο φορέ συνεδριάσει, 7 Ιουλίου και 20 Οκτωβρίου, την περασμένη εβδομάδα δηλαδή με του ηγητέ. Επισκεφθήκαμε τα γραφεία της Frontex στις 30 Σεπτεμβρίου στην Πολωνία, στη Βασοβία. Είχαμε διαβουλεύσει επίσης με τα Εθνικά Κοινοβούλια για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες της αρμοδιότητας ε, της Επιτροπής μας, όπου βέβαια περιλαμβανόταν και η Frontex στις 4 και 5 Οκτωβρίου. Και έτσι φτάσαμε σήμερα εδώ με μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, για να δώσω μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων Τη υπόθεση αυτή, σύντομα όμω για να μπορέσουν να μιλήσουν συνάδελφοι στο μέγιστο δυνατό βαθμό, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καταρχά. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρει πολλού από του συναδέλφου τη Επιτροπής μα, και εμένα βεβαίω, όπω και την ομάδα μου διότι θέλουμε σαφεί εγγυήσει σε αυτόν τον αναθεωρημένο ε, κανονισμό για το σεβασμό από την υπηρεσία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ το θέμα δεν είναι το εάν, αλλά το πώς. Και θα πρέπει να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει απολύτω σοφέ από τι προτάσει τη ότι επιθυμεί μια υπηρεσία υπεράνω πάσα υποψία και άμεμπτη ω προ τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερο κύριο ζήτημα είναι αυτό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ένα περίπλοκο ζήτημα, ένα ζήτημα στο οποίο δεν έχουμε λάβει συγκεκριμένα προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα και για την υπηρεσία της Frontex δηλαδή και κυρίως γιατί η Frontex έχει σήμερα τη δυνατότητα να εξασφαλίζει μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων που διαθέτουν ήδη οι συνοριοφύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχε υπηρεσίες δηλαδή, και τα οποία δεδομένα μπορεί να αξιοποιήσει για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή της ε, λάθρο και παράνομης μετανάστευσης. Ε, δεν μπορεί όμως να επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά. Άρα τι είναι άχρηστα. Και είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα στο αυστηρό, υπογραμμίζω, πλαίσιο της λαθρο και παρανομης μεταναστευσης δεν μπορει ομως να επεξεργαστει τα δεδομενα αυτα αρα τη ειναι αχρηστα και ειναι πολυ λυπηρο το γεγονος οτι η υπηρεσια σε ευρωπαικο επιπεδο δεν ειναι σε θεση να επεξεργαστει προσωπικα δεδομενα στο αυστηρο υπογραμμιζω πλαισιο της. Η πρότασή μου εδώ είναι να αναζητήσω μαζί σας μία διατύπωση που θα επέτρεπε μέσα από μία παράγραφο στην ε, υπηρεσία να ε, χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, φυσικά με όλους τους περιορισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τρίτον, η δυνατότητα κοινή χρήση ανθρωπίνων πόρων. Και εδώ έχω να επισημάνω, Πρόεδρε, ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η χρονική στιγμή ο χρονισμό τη πρόταση την οποία συζητούμε, γιατί έχουμε μια χώρα μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα δηλαδή, η οποία έχει ζητήσει την ανάπτυξη της ε, ομάδας ταχείας αντίδρασης της ε, Frontex ε, και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πρώτη δε φορά αυτό το Σαββατοκύριακο κατέθεσαν έτοιμα για την αξιοποίηση, για την ανάπτυξη μάλλον της Ράπιτες της Frontex οι ελληνικές αρχές. Είναι πολύ θετική εξέλιξη. Πιστεύω το Κοινοβούλιο πρέπει από κάθε πλευρά του να υποστηρίξει την πρόταση αυτή, γιατί το Κοινοβούλιο πριν από τρία χρόνια ήταν εκείνο το οποίο είχε ζητήσει την τροποποίηση τη ε, αρχική ή τη γενική μάλλον ε, νομοθεσία, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η μονάδα η Rabbits. Ε, και είναι η πρώτη φορά, όπω έλεγα, που έχουμε την πιθανότητα ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με την πρόταση είναι και να διευθετήσουμε τις λεπτομέρειες της ε, χρήσης και της λειτουργίας της Rabbits, αλλά και να ε, αναφερθούμε στις άλλες ομάδες, λεγόμενες Frontex Joint Support Teams, τις υποστήριξη δηλαδή. Επίσης, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτραπεί στη Frontex ε, να αγοράζει, εκμισθώνει, χρησιμοποιεί ακίνητα ανάλογα με τις ανάγκες της, ε, πράγμα βέβαια το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάλογα με το αν πρόκειται για αγορά ή εκμίσθωση. Ή εμίσθωση, συγγνώμη. Ε, και φυσικά η αγορά έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στον προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς το να δοθεί η άδεια για αγορά από την υπηρεσία. Γι' αυτό θεωρώ πολύ πιο λογικό, τουλάχιστον στην παρούσα χρονική στιγμή, να δοθεί η δυνατότητα της μίσθωσης μόνο, αλλά βεβαίω δεν θέλω να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων. Άλλα θέματα, πολύ σύντομα. Η διεθνή συνεργασία είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει αρκετού συναδέλφου στην Επιτροπή μα, όπω είναι άλλωστε και το ζήτημα τη βελτίωση των Joint Return Operations. Αυτά και ελπίζω να μπόρεσα να σας δώσω μια καλή επισκόπηση των κύριων σημείων ε, ε, που έχουμε να συζητήσουμε τώρα. Είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα και λόγω τη χρονική τιμή που έχουμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου και του κοιόδους βεβαίως αλλά όλου του συναδέλφου τη Επιτροπή, χάρη στου οποίου πιστεύω μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πουσούτσιλ. Συμβούλιο παρακαλώ. Ράιν, παρακαλώ. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι προβουλευτέ, η ενίσχυση του ρόλου της Frontex είναι πολύ βασικό και προτεραιότητα για το Συμβούλιο. Αυτό έχει φανεί σε πολλά από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στο τελευταίο της 25ης Φεβρουαρίου του 2010, όπου αναφέρονται διάφορα μέτρα για την προστασία των εξωτερικών συμφόρων, συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Από την αρχή της χρονιάς και η Ισπανική Προεδρία και η Βελγική Προεδρία έχει βάλει το θέμα πολλές φορές στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και κάθε μήνα ε, συζητάμε την πρόταση αυτή της Επιτροπής. Συνολικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι αντιπροσωπείες ε, συμφωνούν με την πρόταση της Επιτροπής. Υπάρχουν βέβαια κάποια στοιχεία τα οποία οδηγούν σε συζητήσεις, αλλά στόχος της Προεδρίας και ρόλος της Προεδρίας είναι να φροντίσει να υπάρξει πλήρης προσέγγιση απόψεων. Καταλήξαμε λοιπόν στην προετοιμασία του έργου, στο ότι θέλουμε να έχουμε τις ε, αντιδράσεις κάθε πλευράς. Θέλουμε να φροντίσουμε να υπάρχει μια νομοθεσία με την οποία να συμφωνούν όλοι. Η Προεδρία μας συνεργάζεται με τον κύριο Πουσάτελ που είναι ο εισηγητής σας για την υπόθεση αυτή, αλλά και με τους σκιώδεις εισηγητές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ποιος θα λάβει το λόγο, κύριε Νίλσεν. Κύριε Τέμερμαν, παρακαλώ. Κύριο Τέμερμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όπως γνωρίζετε, ήδη εξήγησε η Επιτροπή Επιτροπή, τις κύριες γραμμές αυτής της πρότασης της, στην Επιτροπή σας εδώ και αρκετό καιρό, ως εκ τούτου δεν πρόκειται να επαναλάβω την ε, κατάσταση συνολικά. Απλώς ήθελα να επισημάνω ορισμένες παρατηρήσεις του εισηγητή στην αρχική του παρέμβαση. ιδιαίτερα με την ενίσχυση τη πτυχή των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων μέσα από την πρόταση αυτή. Η Επιτροπή θέλει να υπογραμμίσει για άλλη μια φορά πω επιδιώκουμε την βέλτιστη δυνατή ισορρόπηση μεταξύ τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών Αφενό μέσω των ε, δραστηριοτήτων τη Υπηρεσία Frontex, του συντονισμού μάλλον, και αφετέρου τη λειτουργική ικανότητα δράσης της ίδιας της υπηρεσίας, δηλαδή να μην ε, ε, ε, παρεμποδίσουμε ουσιαστικά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Επιδιώκουμε λοιπόν σε συνεργασία με τους ε, εταίρους μας στην υπόθεση αυτή να εξασφαλίσουμε αυτή την ε, ισορροπία. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Το ανέφερε και ο εισηγητής πως δεν αποτελεί αντικείμενο της προτάσεως της Επιτροπής. Διότι θέλησαμε πρώτα να εξασφαλίσουμε μια επισκόπηση των διαφορών θεμάτων που είχαν σχέση με τη συλλογική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις ε, υπηρεσίες GHA ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή των συνόρων. Ε, και ως εκ τούτου τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού έκανε αυτή την επισκόπηση, εξετάζει το θέμα και θα πρέπει σε μεταγενέστερο στάδιο να υποβάλουμε νέα πρόταση για την υπόθεση αυτή. Για την κοινή χρήση ανθρώπινων πόρων. Είτε πρόκειται για τους ανθρώπινους αλλά ακόμα και για τους τεχνικούς ε, πόρους, θα ήθελα να δώσω μια διαφορετική προοπτική, ιδιαίτερα όσον αφορά τη τεχνική σκοπιά. Μια μελέτη σκοπιμότητας που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στη Frontex εξετάζει τον καταλληλότερο τρόπο, δηλαδή τη δυνατότητα αγοράς ελαφρότερου υλικού ή μίσθωσης βαρύτερου υλικού πρόθεση της πρώτας επιτροπής δεν είναι ξαφνικά αυτή η υπηρεσία να αναλάβει όλο το υλικό, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, που τις διαθέτουν τα κράτη-μέλη κατά, κυριαρχία κατά ιδιότητα, κατά ιδιοκτησία, συγγνώμη. Δεν θέλει δηλαδή να βρεθεί η Frontex να αγοράζει τρία ή τέσσερα μεγάλα σκάφη, σκάφη του λιμενικού, ακτεωρούς ε, ή οτιδήποτε άλλο μεγάλο ε, μηχάνημα ή εξοπλισμό. Κοιτάμε περισσότερο με τι είναι σκοπιμότερο και τι εξασφαλίσει την περισσότερη προσθέμενη αξία. Και αυτά βέβαια πάλι σε, συνδυασμό και με τα θέματα που θέτει ο εισηγητή για τη διεθνή συνεργασία και την ε, υποχρέωση παρακολούθησης του κώδικα ε, χάρη στον οποίο νομίζω εξασφαλίσουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης από πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και την έκθεση αλλά και τη συζήτηση γενικότερα του θέματος αυτού με την ε, ελπίδα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μια καλή και στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έτσι ώστε να διεκπαιρεώσουμε το θέμα αυτό εν χρόνο. Ευχαριστώ, λίγο Και τώρα Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Λαπρινίδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο Σάιμον σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με το Frontex και θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει να βρούμε ένα σωστό τρόπο να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Να πω καταρχάς ότι πράγματι η Ελλάδα ζήτησε από την δύναμη ταχείας ανάπτυξης η κατάσταση στα βόρεια σύνορά μας με την Τουρκία είναι πλέον ανυπόφορη το 85% περίπου των παράνομων μεταναστών που μπαίνουν ε, στην Ελλάδα μπαίνουν από τα σύνορα με την Τουρκία. Η κατάσταση είναι εκτός ολέγχου και πράγματι η θετική απάντηση της Frontex ήταν καλοδεχούμενη. Θα ήταν καλό να υπάρξει βελτιωμένη συνεργασία με την Τουρκία στο συγκεκριμένο αυτό επί τη βάση ε, της συνεργασίας του Frontex και της Τουρκίας. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να βάλουμε στην έκθεση το εξής. Αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι κυρίως λειτουργικές. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση ε, να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνει το Frontex και όχι να χρησιμοποιήσουμε τις συμφωνίες αυτές για άλλα θέματα. Το λέω αυτό γιατί σε κάποιες από τις διαπραγματεύσεις η Τουρκία προσπαθεί να διαπραγματευτεί ουσιαστικά, να κάνει παζάρια θα έλεγα, με το θέμα αυτό, με άλλα θέματα, οι διεκδικήσεις τις οποίες θεωρεί ότι έχει και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Θα πρέπει λοιπόν ε, να πατήσουμε και στις συμφωνίες τις αντίστοιχες που έχουμε με άλλες χώρες και το ίδιο να κάνουμε με την Τουρκία. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα στην υπηρεσία και τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για το ξεκίνημα της προσπάθειας αυτής, αλλά και τον τερματισμό. Η Frontex μπορεί να τερματίσει τη δραστηριότητά της πληροφορώντας για κάποιους λόγους την συγκεκριμένη χώρα. Είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία την οποία θέλουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια συνεργασία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στήριξης και η απότομη διακοπή μιας τέτοιας προσπάθειας επιχείρησης δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από σαλήνη. Σάιμον, αυτό είναι ίσως ένας από τους λόγους που θα πρέπει το Frontex να έχει κάποιο εξοπλισμό ο οποίος να είναι αποκλειστικά για αυτόν δικός του και όχι να υπάρχει μια κάποια χώρα η οποία προσφέρει το υλικό και αποφασίζει ότι α, δεν μπορώ πια να το προσφέρω γιατί πρέπει να το στρέψω αλλού. Και εξαρτάται αυτό και από το αν θα χρησιμοποιηθεί το Frontex περισσότερο. Ε, σε αυτή την περίπτωση ε, η συνεχής χρήση των υλικών αυτών και των εξοπλισμών από τρίτες χώρες μπορεί να είναι κάτι το όχι ιδιαίτερα σίγουρο και βέβαιο και θα πρέπει εν πάση περιπτώσει όλα αυτά να τα καλύψουμε. Τέλος να πω ότι σε κάποια φάση στο κείμενο υπάρχει μια προβληματική αναφορά στις θαλάσσιες επιχειρήσεις και ότι το Frontex θα καθορίζει ποιες είναι οι νομικές ε, ρυθμίσεις ε, στα πλαίσια της, των θαλασσίων επιχειρήσεων. Όλους μας αφορούν, είπαμε, οι νομικές αυτές ρυθμίσεις. Εμείς θα πρέπει να μην υποκαταστήσουμε το Frontex, αλλά καλό θα είναι αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση να τη διευκρινίσουμε, γιατί δημιουργεί συγχύσεις και να πούμε ότι ο νόμος ο οποίος θα εφαρμόζεται είναι ο ισχύων και θα πρέπει να γίνεται σεβαστός και να εφαρμόζεται χωρίς καμία άλλη ε, απόκληση από τη γραμμή αυτή. Κυρία Βίξτρομ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Σάιμον γιατί κάλυψε τις ανησυχίες μας και τις προτάσεις που του κάναμε ήδη από την αρχή της διαδικασίας. Είναι προφανές ότι το Frontex χρειάζεται μια πιο ξεκάθαρη εντολή. Όλοι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας λοιπόν. Και εγώ ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί οι ομάδες αυτές ε, ε, ανάπτυξης που δημιουργήθηκαν το 2000 λεπτά κινητοποιήθηκαν για πρώτη φορά και αυτό δείχνει την μεγάλη σημασία την οποία έχει το Frontex και θα έχει στο μέλλον και βλέπουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ωφεληθεί πλήρως από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μιλάμε συνεχώς για την αλληλεγγύη, αλλά τώρα την δείχνουμε στα πλαίσια της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Όλοι λοιπόν θα πρέπει τώρα να μπορούν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπως αυτές αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία θα ήθελα να επιμείνω περισσότερο. Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες, σαν παράδειγμα. Οι συμφωνίες αυτές δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο έγκρισης από το Κοινοβούλιο, όπως άλλες διεθνείς συμφωνίες, γιατί το Φρόντες χαρακτηρίζεται από μια κάποια αυτονομία. Αλλά να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται για όλες τις μορφές ε, διεθνούς συνεργασίας τις οποίες εμπλέκεται το Frontex ιδιαίτερα με αρχές τρίτων χωρών. Είναι πολύ σημαντικό και ίσως να γίνει ακόμα πιο σημαντικό όταν η κατάσταση ε, αλλάξει. Σχετικά με την αγορά ή τη μίσθωση του εξοπλισμού κτλ. Αυτή η συζήτηση Ε, δεν είναι ίσως ε, τόσο ασήμαντη γιατί τελικά αυτό το οποίο διαφοροποιεί ε, τους ισχυρούς από τους ασθενείς είναι η ποιότητα των μέσων τα οποία χρησιμοποιούν. Συνεπώς θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όσο μπορούμε τον προϋπολογισμό αλλά με λειτουργικό πάντα τρόπο. Έχει επίσης σημασία η εκπαίδευση των μεθοριακών φρουρών, των συνοριοφυλάκων, ε, να περιλαμβάνει και το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ήδη σιγά σιγά γίνεται ε, στα πλαίσια της Βαρσοβίας, του Frontex και αυτό θα πρέπει να ισχύσει ακόμα περισσότερο στην περίπτωση της ανάπτυξης της ε, συγκεκριμένης αυτής δύναμης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη στις κοινέ επιχειρήσεις και στις, ε, στη συνέχεια των επιχειρήσεων αυτό που έχει σημασία είναι ακριβώς η σταθερότητα και η διασφάλιση της συνέχειας, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι σαν παράδειγμα περνούν από τις διαδικασίες επανεισδοκής, Σαν παράδειγμα έχουν ε, επιστραφεί πίσω χριστιανοί Ιρακινοί στο Ιράκ, τους παρατάμε στο αεροδρόμιο και δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει αυτοί οι άνθρωποι από εκεί και πέρα. Αν στόχος του Frontex είναι να κάνει τέτοιου είδους κοινέ επιχειρήσεις, θα πρέπει να τις κάνει αλλά όντα σίγουροι για το τι συμβαίνει σε αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης. Λοιπόν, αυτές ήταν κάποιες από τις λεπτομέρειες τις οποίες θα ήθελα να σταθώ. Να πω πάντως γενικά συμφωνώ με τον εισηγητή και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ κυρία Βίξον. κυρία Φλότρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια αντίδραση σε σχέση με το αίτημα της Ελλάδας για την ανάπτυξη των ε, μονάδων της Frontex στα σύνορά της. Έχει μια κάποια λογική αυτό. Γιατί, διότι τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι οι μη ομαλές ροές μετανάστευσης που είχε να χειριστεί η Frontex στην νότια αυτή της Μεσογείου έχουν λίγο πολύ αυξηθεί μάλλον όσο μείωσε η Frontex στην νότια όχθη της Μεσογείου τις μεταναστευτικές ροές της παράνομες, τόσο ενισχύθηκε λίγο πολύ, κατά τη στοιχεία δηλαδή, κατά αναλογία, η ροή μεταναστευτική μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Λογικό είναι λοιπόν να στήσει η Ελλάδα από τη Frontex να παρέμβει στα ε, σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία. Από εκεί και πέρα βέβαια το ζήτημα τη αναθεώρησης τη εντολή τη Frontex και το βαθμό στον οποίο οι ε, δράσει και η λειτουργία τη Frontex είναι σύμφωνε με το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν διευκρινίζεται από την ε, πρόταση αναθεωρημένη εντολή και δεν ξέρω γιατί. Ίσως η κατάσταση της Ελλάδας να περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, διότι εν τέλει έχουμε να κάνουμε μια διπλή προσέγγιση εδώ. Δηλαδή είναι πότε ε, διακρατική οργάνωση Frontex που απλώς συντονίζει τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη-μέλη αλλά υπό την ευθύνη όταν πρόκειται για εξωτερικά σύνορα του εμπλεκομένου κράτους μέλους. Η πρόταση που έχει καταθέσει η Ελλάδα κατά την άποψή μου ανοίγει μια νέα προοπτική ευθύνης η αναζήτηση του ποια θα είναι η αρχή αρμόδια για αποζημίωση ενδεχομένω σε περίπτωση ζημίας και από την άλλη όταν ξεκινάει η Frontex κάποια σχέδια και πιλωτικά ακόμη τότε η ο επιμερισμός της ευθύνη σε περίπτωση ζημίας θα μπορούσε να είναι εξ ολοκλήρου σε επίπεδο Frontex. Άρα έχουμε καταλήξει σε ένα φλου τελικά. Ε, έχουμε μία Frontex και μια διακρατική οργάνωση, δηλαδή διατίθεται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια μέσα για διακρατική συνεργασία μεταξύ των κρατών ή αλλιώς η Frontex είναι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία και άρα είναι διαφορετικό το νομικό πλαίσιο στο οποίο δρά. Η πρόταση κατά την άποψή μου μόνο διατηρεί την αμφισημία και μόνο ενισχύει τις δυνατό, το δυναμικό δηλαδή και τις εξουσίες της υπηρεσίας, δηλαδή ενισχύει ουσιαστικά την αμφισημία, την αβεβαιότητα. Και βέβαια μπορώ να αντιληφθώ και να ε, κατανοήσω, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο εισηγητή μα θα μεριμνήσει ιδιαίτερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ε, θεμελιώδει ελευθερίε. Κατανοώ επίση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη ε, για αναθεωρημένη εντολή έχει καταθέσει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε προτάσεις, ε, παραδείγματι κατάρτιση για τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, ε, διαδικασίες επανεισδοχής κτλ. Εδώ έχουμε να κάνουμε θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα στη διεθνή προστασία, το δικαίωμα της μη, της μη αποπομπής σε μια χώρα στην οποία υπάρχει κίνδυνο τα δικαιώματα των ανηλίκων είναι θεμελιωδέστατα όλα αυτά. Πλην όμως τελικά δεν φτάνουμε μέχρι τέλους αυτό το συλλογισμό και τη λογική, διότι δεν υπάρχει ένας ε, ικανός, επαρκής, και οργανωμένος μηχανισμός που να επιτρέψει να παρακολουθούνται συστηματικά αυτά τα ζητήματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και εμείς ως βουλευτές τελικά ε, μόνο όταν ε, θεωρήσει σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερωνόμαστε ή θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε δεχομένως για τέτοια πράγματα. Θα εξαρτώμεθα από την Επιτροπή δηλαδή. Ενώ εμεί θέλουμε να έχουμε μηχανισμούς με ανεξάρτητη εποπτεία και γνωμοσύνες, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλιώ δεν πρόκειται να έχουμε σωστικά αποτελεσματάκια από τι εκθέσει που έχει καταθέσει μέχρι τώρα τουλάχιστον η υπηρεσία αυτή. Διαπιστώνεται ότι είναι πολύ μεγάλη δυσκολία ε, ε, του σεβασμού των δικαιωμάτων. Βεβαίω θα γίνουν οι καταρτήσει, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε και ένα μηχανισμό κατάρτιση, αξιολόγηση, ενδεχομένω και διερεύνηση ε, του επιμερισμού τη ευθύνη σε περίπτωση ζημία. Γιατί πάντω θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εξασφαλίζουμε την προστασία των δικαιωμάτων, την ουσιαστική προστασία, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα της αποκατάστασης ή της αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας. Έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται ποτέ αυτές οι παραβιάσεις. Και εμείς ως βουλευτές πρέπει να ενημερωνόμαστε τακτικά για τις δραστηριότητες και την αξιολόγησή τους, τη σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά άλλωστε μας έχει εμπνεύσει και η έκθεση της Επιτροπής των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων και ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην κυρία Λόκμπιντερ που είναι εδώ δίπλα και ακούει, παρακολουθεί τις ε, ε, συζητήσεις μας. Φαντάζομαι ότι θα λάβει υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις. Πάντως πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για να έχουμε ουσιαστική ε, προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι έχουμε πολλή δουλειά Γι' αυτό ας σταματήσουμε με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε ένα ακόμα θέμα πριν διακόψουμε στις 12.30. Οπότε να μπορέσουμε μετά να ξαναρχίσουμε στις 3, έτσι όπως προβλέπετε από την ημερήσια διάταξη. Κλείνει λοιπόν ο κατάλογος. Προτείνω να πάρουν το λόγο ακόμα η εξή, αλλά για λίγο. Η κυρία Γκυγιόμ πρώτα. Μη μακρηγορείτε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ είχα καταλάβει στην πρόταση της Επιτροπής, μπορεί βέβαια να κάνω και λάθος, ότι μιλάμε για μια διπλή ισορροπία. Από τη μια αυτονομία του οργανισμού και από την άλλη ότι αποτελεί ένα μέσο που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η μία ισορροπία. Και από την άλλη ισορροπία ανάμεσα σε μια προσέγγιση υπέρ της ασφάλειας, αλλά από την άλλη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ έτσι το είχα καταλάβει. Γιατί εγώ θέλω να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Και δεν ξέρω κατά πόσο την έχουμε πετύχει. Φαντάζομαι ότι δεν είμαι μόνο εγώ που νιώθω άβολα, γιατί δεν αισθάνομαι ότι έχουμε μια πλήρη άποψη για τις δραστηριότητες της Frontex. Στη Βασοβία η επίσκεψή μας ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα, όμως δεν κατάφερε να μας καθησυχάσει πλήρως. Τέσσερα σημεία, μια που με ζητάτε να είμαστε σύντομοι. Αλλά δεν είναι και τα μόνα που θα είχα, αλλά που θα έπρεπε οπωσδήποτε να κοιτάξουμε και να μελετήσουμε. Πρώτα απ' όλα για τον ρόλο του οργανισμού και των κρατών μελών. Οι μετανάστες δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και έχω την εντύπωση ότι παίζουν κρυφτούλοι οι Frontex με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θέλουν να έχει την ευθύνη η Frontex, απ' την άλλη μεριά ο οργανισμός συντονίζει και κρύβεται πίσω από αυτό το συντονιστικό ρόλο. Δεύτερον, κάτι άλλο. Ε, θέλουμε μια Ευρώπη που να προστατεύει. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη ότι η δημιουργία οργανισμών για τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ένας ανεξάρτητος έλεγχος για την αναγκαστική επιστροφή μπορεί να διασφαλίσει την αξιοπρεπή μεταχείριση των μεταναστών. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προβλέψουμε ένα σύστημα εποπτείας και ελέγχου για όλες τις δραστηριότητες της Frontex. Τρίτον, αναφέρθηκε και αυτό λίγο, να λειτουργεί με περισσότερη διαφάνεια η Frontex. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές λάβαμε έκθεση δραστηριοτήτων ρητορικού χαρακτήρα με ένα σωρό στατιστικά στοιχεία. Δεν μαθαίνουμε όμως τίποτα για την ποιότητα του έργου της Frontex. Καλό θα ήταν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται καλύτερα όσον αφορά τις δραστηριότητε της Frontex και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που κάνει με τρίτες χώρες. Τέλος, παρόλο που η διάσταση είναι ε, μεγάλη και το ξέρουν και ο συγητής ε, και οι σκιώδεις, αλλά θα είμαι σύντομη, προσοχή στα προσωπικά δεδομένα. Χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνες. Δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά σε αυτό. Για να δούμε ποια θα είναι η μεταχείριση που επιφυλάσσει η Frontex στα προσωπικά δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με την Europol όσον αφορά τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η Frontex. Στο στάδιο αυτό λοιπόν η πρόταση είναι σημαντική, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να την ξανασυζητήσουμε και να ξανασυζητήσουμε γενικότερα τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε τι νόημα δίνουμε στην διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα των προσωπικών δεδομένων συμφωνώ θα πρέπει όμως να μην επικαλύψουμε αυτά τα οποία ήδη κάνει η Ευρωπόλ. Όταν δίδουμε νέες αποστολές στο Frontex σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, σαν παράδειγμα. Ήδη βέβαια το Frontex επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ιδιαίτερα για τις διαδικασίες της επανεισδοχής. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ασχολούμεθα με το θέμα αυτό. εφόσον έχουμε, επαναλαμβάνω, στη διάθεσή μας δομές οι οποίες εκπληρούν α, ε, τις επιθυμίες μας. Τώρα, φυσικά για τα θέματα των παζαριών και της διαπραγμάτευσης, εδώ τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο ούτε το ενός ούτε το άλλο. για την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Και στα πλαίσια της επίσκεψής μας στη Βαρσοβία ακούσαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν δέχονται τις ε, υπηρεσίες τους εύκολα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα χωρίς το Frontex. Τώρα εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί που ξοδεύουμε τα χρήματά μας να δημιουργούν προστιθέμενη αξία οι δαπάνες. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι να βελτιώσει το σύστημα χορήγησης ασύλου και ίσως οι προσπάθειες μας θα πρέπει να είναι περισσότερο εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς που αιτούνται ασύλου. Πολλοί από αυτούς ε, που πηγαίνουν στην Ελλάδα θέλουν να ζητήσουν άσυλο, έχουν δικαίωμα να το κάνουν σύμφωνα με τους κοινοτικού κανόνες, αλλά δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά οι κανόνες αυτές, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες εκεί και δεν νομίζω ότι ο έλεγχος των συνόρων είναι, ε, θα έλεγα, η λύση στο πρόβλημα. Το Frontex είναι στην ουσία σύνοριοφύλακες, δεν είναι ε, άνθρωποι που ελέγχουν τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Στα πλαίσια των συμφωνιών με τρίτες χώρες και στα πλαίσια των τακτικών ε, κοινών επιχειρήσεων υπάρχει ένας φαιός χώρος ανάμεσα στο τι είναι λειτουργικό και στο τι είναι πολιτικό το Frontex θα πρέπει να προσέξει και αυτό τις δραστηριότητές του και θα πρέπει και εμείς να ελέγχουμε ακριβώς το λειτουργικά είναι, ε, το ποια στοιχεία της λειτουργίας ακριβώς του Frontex δεν είναι πολιτικά. Δεν έχω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Ένστ. Κυρία Ένστ. Καινούριο αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πολύ καλό, πιστεύω, το να εμπλακούμε σε κάθε βήμα αυτή τη διαδικασία και να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το περίπλοκο ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Για διάφορα σημεία, λοιπόν, έχω κάποιε παρατηρήσει. Πρώτη ερώτηση και κύρια πρέπει να αναλογιστούμε τι ακριβώς επιδιώκουμε με το Frontex, τι θα προκύψει εν τέλει από την δραστηριοποίησή της. Θα είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων, με τον έλεγχο της διάβασης των συνόρων, με την επικτήρηση των συνόρων, με την παρεμπόδιση της παράνομης μετανάστευσης, λαθρομετανάστευσης, εν τέλει δηλαδή μια σκοπιά ασφάλειας αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε εμείς εάν θέλουμε να είναι αυτόνομη η Frontex ή όχι. Και αν δεν θέλουμε να είναι αυτόνομη, συγκεκριμένα τι ρυθμίσεις θέλουμε να επιβάλλουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε κάθε ζήτημα και σε κάθε θέμα συγκεκριμένα, έτσι ώστε να μην υπάρξει αυτονομία, αυτόνομη δράση, αυτοδιαχείριση, και πιστεύω ότι εμεί ω βουλευτέ είναι απαραίτητο ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλεκόμαστε σε κάθε διαδικασία. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Είναι ζωτική σημασία επίση και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να εμπλέκονται σε κάθε στάδιο, φερειπίν στην ανάλυση κινδύνου. Πώ είναι δυνατόν να γίνει η ανάλυση κινδύνου χωρί συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων η οποία βέβαια έχει και πολύ μεγάλη σημασία στη νέα αυτή ε, διαμόρφωση τη εντολή τη Frontex. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε για άλλη μια φορά και όχι ε, σε γενικού όρου, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Δεύτερον, ε, ουσιαστική επιδίωξη και εν τέλει ο πυρήνα των συζητήσεων μα από εδώ και μπρο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδη ελευθερία. Ε, και πιστεύω ότι μέλημα ιδιαίτερα τη δική μα ομάδα οπωσδήποτε, αλλά όλων θα πρέπει να είναι το να εξασφαλίσουμε σε σχέση με την φρόντιση ε, την ουσιαστική διαφύλαξη των αρχών του ασύλου, την ουσιαστική παροχή δικαιώματος ασύλου όσο το χρειάζονται, ατομικά. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Και πώς θα το ε, αντιμετωπίσουμε με δεδομένο το σχετισμό με τη λεγόμενη λάθρο μετανάστευση. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά και σε λεπτομέρεια με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν δεν εδρεωθούν αυτά, αν δεν προστατευτούν ικανοποιητικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τρίτη παρατήρηση, έχω πολύ σοβαρές ανησυχίες, πολύ σοβαρές ανησυχίες ως προς την συνεργασία με τρίτα κράτη, όπως λέγεται. Όταν πρόκειται ιδιαίτερα για τρίτα κράτη τα οποία δεν έχουν λαμπρές επιδόσεις στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η συνεργασία, εδώ είμαι πολύ επιφυλακτική όπως λέω. Τέταρτο σημείο, επιφυλάξεις πολλές έχουν διατυπωθεί, άλλωστε και από τον ε, εκπρόσωπο για, τα, για την προσέγγιση προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συναντήσουμε Τετάρτη, ε, ως προς την διαχείριση των δεδομένων ε, που συλλέγει η Frontex από δραστηριότητές της και ε, υπάρχει ο κίνδυνος να μας ξεφύγει η κατάσταση και να μπορούμε πλέον να την ελέγξουμε. Επίσης, ο αρμόδιο, ο υπατός εκπρόσωπος για, ανθρώπινα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα μας ε, πει, πιστεύω, σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν η Frontex να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ε, και να τα διαθέτει. Αυτό είναι κάτι το οποίο ασφαλώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στι περαιτέρω συζητήσει και τι διαπραγματεύσει για την διαμόρφωση τη εντολή τη Frontex. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπα-Νικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εντάχει και προσπαθώντας να συμπληρώσω στα όσα υπόθηκαν και να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, προσθέτω και εγώ τα εξή. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την αναφορά που κάνουν στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι αυτή η συζήτηση αφορά την Ελλάδα καθώς η ίδια η Frontex, κυρίως στην Ελλάδα, καθώς η ίδια η Frontex αναφέρει ότι το 80 με 85% των ε, ανθρώπων εκείνων που παράνομα προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρώπη το κάνουν από την Ελλάδα. Και πράγματι αντιμετωπίσαμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ μεγάλη πίεση και αποτελεί βεβαίως ένα γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί και έκτακτο και γι' αυτό είναι σημαντική η ανταπόκριση που είχαμε από τη Frontex και από την Επιτροπή, από την κυρία Μάλστρομ στο αίτημα της Ελλάδας αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς πλέον επειδή για να γίνει αντιληπτό αυτό για τους συναδέλφους επειδή στο Αιγαίο η παρουσία και της Frontex και των ελληνικών δυνάμεων βελτιώνεται και είναι πιο επικίνδυνη η μετακίνησή τους με τους διαφόρους που προσπαθούν να επιτελέσουν τέτοιους σκοπούς, πλέον εκείνοι που παράνομα προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη δεν επιλέγουν την είσοδο μέσα από τη θάλασσα, αλλά πηγαίνουν ψηλά στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας μέσω της Τουρκίας και από εκεί χερσαία προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα. Και γι' αυτό εκεί η κατάσταση ήταν δραματική και είναι δραματική και η ανταπόκριση είναι πολύ σημαντική. Βεβαίως όταν αναφερόμαστε στο θέμα της έμπρακτης αλληλεγγύης που πρέπει να δείχνουμε για τα θέματα αυτά της λαθρομετανάστευσης είναι ε, πολύ σημαντική η συζήτηση ε, για την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση της Frontex, ενός οργανισμού που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια να λειτουργεί και η δική μας θέση είναι ότι με την παρουσία του συνδράμει καθοριστικά στην καταπολέμηση του φαινομένου. Τρεις τεχνικές παρατηρήσεις αναφέρθηκαν ήδη, επιγραμματικά λέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τις τρίτες χώρες να εστιάζουμε αποκλειστικά σε τεχνικά θέματα και να μην έχουμε εμπλοκή άλλων παραμέτρων. Ε, δεν είναι τυχαίο που μέχρι τώρα δεν έχει υπογραφεί τελικά η συμφωνία της Τουρκίας με τη Frontex, όπως δεν έχει υπογράψει επίσης η Τουρκία τις συμφωνίες επανεισδοχής των ε, παράνομων μεταναστών για την Ευρώπη. Κάθε φορά η κυρία Μάλστρομ όταν μας ενημερώνει μας λέει ότι βρισκόμαστε σε τελική φάση, ακόμη όμως δεν έχουμε κύριε Πρόεδρε τελειώνω, δεν έχουμε ακόμα ε, συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι επίσης σημαντικό όταν η Frontex τερματίζει κάποια ε, επιχείρηση αυτό να γίνεται σε συνεννόηση με το κράτος μέλος υποδοχής όπως επίσης ίσως θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε και αυτό ε, θα βρω κάποια ευκαιρία να το συζητήσω και με τον εισηγητή μας τον κύριο Μπουζουτήλ τον, οποίο και ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια το ζήτημα της περαιτέρω χρηματοδότησης των κινήτρων που θα μπορούσαν να δοθούν σε σχέση με τον εξοπλισμό που θα μπορούσαν να διαθέτουν τα κράτη-μέλη πέρα του ελαχίστου όπως προβλέπεται στο κείμενο που έχουμε μέχρι τώρα. Ε, επιφυλάσσομαι για, για την ε, περαιτέρω συζήτηση, κλείνοντας μόνο μία φράση για τα θέματα του ασύλου. Βεβαίως η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει και δέχεται πολύ μεγάλη πίεση στα θέματα αυτά και έχει σημαντικές αδυναμίες. Πρέπει να θυμόμαστε όμως όλοι ότι για να λύσουμε και αυτά τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις τεράστιες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε λόγω του Δουβλίνο 2, που είπαμε ότι μπορεί να ανασταλεί, τελικά όμως αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει πάνω απ' όλα να προσπαθήσουμε να περιφρουρήσουμε τα σύνορα της Ευρώπης ξεκινώντα κανεί να φυλάει σωστά τα σύνορά του, από εκεί και πέρα μπορεί να δρομολογήσει και τη διαχείριση όλων των άλλων πολύ σημαντικών ζητημάτων, όπως αυτά που αφορούν τα θέματα του ασύλου. Σας ευχαριστώ και επιφυλάσσουμε βεβαίως για τις επόμενες συζητήσεις. Thank you. very much and... Uh, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ Σάιμον για τις προσπάθειες που έχει κάνει να βελτιωθούν οι εργασίες της Frontex. Είναι πραγματικά πολύ υπεύθυνο από πλευρά μας. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ λιγάκι στο θέμα της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν όντω πολλοί λαθρομεστανάστες που προσπαθούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ επιστρέφω από τα Δυτικά Βαλκάνια και πρέπει να ξέρουμε ότι ο αριθμός των λαθρομεταναστών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και στην Σερβία και την Μακεδονία, λέει μιλήτρια. Πώς λοιπόν θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ξέρετε ότι για αυτές οι χώρες είναι πιο φτωχές και εκεί οι κυβερνήσεις χρειάζονται μεγάλη στήριξη. Ξέρετε επίσης ότι η αστυνομία δεν συνεργάζεται καλά. Γιατί, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορούν να προσφέρουν άσυλο, καλές συνθήκες, ούτε και στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι από διάφορα κανάλια τελικά περνάνε και φτάνουν και στη Σερβία και στη Μακεδονία και στο Πέδιο. Οι χώρες αυτές οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Μιλάμε για την ανάπτυξη δύναμης, είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα βέβαια, αλλά να λάβουμε υπόψη μας εδώ και τις άλλες χώρες που και αυτές θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή και να φροντίσουμε να τις στηρίξουμε και αυτές. Τώρα έρχομαι στα άλλα θέματα τα οποία έθεσε ο Σάιμον για την Frontex. Την επεξεργασία δεδομένων, για παράδειγμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τον οργανισμό, για τη Frontex. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορεί υπεύθυνα να επεξεργάζεται τα δεδομένα η Frontex. Συγχρόνως όμως είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε και αυτό που είπες εσύ, δηλαδή τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να υπάρχουν ξεκάθαρες εγγύσεις ότι ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχομαι τώρα και σε ένα άλλο θέμα στο θέμα των περιουσιακών στοιχείων. Δεν ξέρω αν ξέρουμε τελικά πού πηγαίνουν ακριβώς τα χρήματα και πώς δαπανώνται. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται επί Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην Frontex και την χώρα στην οποία βρίσκεται η Frontex. Όπως είπε και ο Σταύρος, η συνεργασία αυτή με τα κράτη-μέλη η συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, ποιο εξοπλισμό είναι καλύτερο, που μπορεί να διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Εξαρτάται από την κατάσταση επιτόπου ποιο είναι ο καλύτερο εξοπλισμό. Γι' αυτό πιο συχνά θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν για να ξέρουμε πώς μπορούμε καλύτερα και να αντιδράσουμε με που έχουμε σήμερα τη συζήτηση αυτή για το έργο της Frontex και για το τι γίνεται επί τόπου. Ελπίζω ότι θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ και εγώ τον Σάιμον Μπουσάτελ για τη δουλειά του και γιατί έχει πραγματικά ανοιχτό πνεύμα. Είμαι σίγουρη ότι θα φροντίσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα τα συμπεριλάβει επαρκώ στην εκθεσή του, γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για τον οργανισμό αυτό, λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα ευτυχή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα υποβάλλει αυτή την πρόταση. Είναι ένα νέο οργανισμό. Και επειδή ήμουνα πέρυσι εισηγήτρια για την απαλλαγή, Πρέπει να σα πω ότι τα τελευταία χρόνια ζητήσαμε πολλά από αυτόν τον οργανισμό, παρόλο που δεν ήταν πάντα καλά έτοιμο και προσαρμοσμένο για την αποστολή του. Καλό είναι λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα κοιτάει την ανανέωση της εντολής. Πράγματι τα τελευταία χρόνια πήγαν πολλές πιστώσεις εκεί. Και ίσως ο οργανισμός ξεπεράστηκε λιγάκι από τα γεγονότα. Είναι πολύ καλό νέο λοιπόν η μεταρρύθμιση της εντολής. Οι σημαντικές αποστολές για τη διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων μας, και οι προσωπικές ε, εγγύσεις για τα δεδομένα είναι τα δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να προωθήσουμε. Θέλω όμως πάντως να φροντίσουμε να μην ε, επιβαρύνουμε πολύ τις διαδικασίες. Όπως σας είπα, ξεπεράστηκε ο οργανισμός από το όσα ζητήσαμε. Ήταν ένας νέος οργανισμός και βέβαια δυσκολεύτηκε. Πρέπει να έχουμε περισσότερο προσωπικό στη Frontex, πρέπει η εντολή της ε, της Frontex να είναι κάτι ξεκάθαρο, να ξέρουμε ποιος κάνει τι και διευθυντής. Μερικές φορές δεν υπήρχε αρκετός διάλογος ανάμεσα στα κράτη-μέλη και το προσωπικό του οργανισμού. Πρέπει και αυτό να είναι ξεκάθαρο γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για τη μεταρρύθμιση της εντολής της Frontex. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπρόγκς τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του Frontex περιορίζεται από την έλλειψη προσωπικού. Ε, η ανάπτυξη των δυνάμεων του Frontex στην νοτιοδυτική Ευρώπη μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στην ε, νέα ανάπτυξή του στα σύνορα με την Τουρκία μήπως θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιήσουν ε, και κάποιες χώρες το προσωπικό που έχουν στη διάθεσή τους ε, για να συμπληρώσουν τις αποστολές του Frontex. Τι νόημα έχει να τρέχουν και να κάνουν άσχετους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, να προγραμματίζουν άχρηστους πολέμους στο Ιράν και να μην μπορούν να προστατεύσουν τα σύνορά τους. Το πρόβλημα με τους, με αυτούς που ζητούν άσυλο είναι πολύ σύνθετο. Αυτοί οι οποίοι είναι γνήσιοι ε, πολίτες οι οποίοι ζητούν άσυλο πρέπει να στηριχθούν, αλλά όχι οι υπόλοιποι που στην ουσία είναι τμήμα της οικονομικής μετανάστευσης. Μετά από αυτήν την ανταλλαγή απόψεων επιστρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και στο τέλος τον Μπουσουτήλ, τον εισηγητή μας. Λοιπόν, θα ήθελε το Συμβούλιο ή η Επιτροπή να κάνουν κάποια σχόλια σχετικά με αυτά τα οποία ακούστηκαν. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Σύντομα, Πρόεδρε, για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση, όταν αναφερθήκαμε στο θέμα των, στην ισορροπία ανάμεσα στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην λειτουργική ε, πρακτική την οποία ακολουθούν τα Frontex, το Frontex, είναι σαφές ότι εμείς δεν είμαστε το κατάλληλο σώμα για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στα δύο, απλά λέμε ότι ο κανονισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις και θέλουμε οι διαδικασίες αυτές που θα εφαρμοστούν να καταστήσουν δυνατό για την υπηρεσία Frontex να λειτουργήσει με τον σωστό τρόπο. Μετά από αυτά τα οποία άκουσα στην συζήτηση μέχρι τώρα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα-δύο από αυτά τα στοιχεία που ακούστηκαν όπου απαιτείται νομίζω μια κάποια μεγαλύτερη ευκρίνεια. Πρώτον, και αυτό είναι το σημείο αφετηρίας αν θέλετε, εμείς στα πλαίσια αυτής της πρότασης δεν δημιουργούμε ε, μια ανεξάρτητη υπηρεσία Frontex και όταν λέω ανεξάρτητη εννοώ ότι ο έλεγχος των πολιτών στα εξωτερικά σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ως έχει, είναι πλήρης δηλαδή η ευθύνη των κρατών μελών. Όχι το επειδή η υπηρεσία αυτή θα έχει κάποιο εξοπλισμό στη διάθεσή της, θα αλλάξει και η ευθύνη της και η αποστολή της. Αυτό είναι το πρώτο σημείο διευκρίνησης. Το δεύτερο σημείο. Εννοείται ότι όταν το Frontex ξεκινά κάποιες διαδικασίες και άκουσα και για τον τερματισμό των κοινών ε, αυτών επιχειρήσεων, είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις αυτές ε, διεξάγονται σε πολύ στενή συνεργασία με την χώρα που φιλοξενεί τη δύναμη του Frontex. Και ο τερματισμός ε, των επιχειρήσεων αυτών θα πρέπει να υπόκειται στις ίδιες γραμμές, όχι ότι ξαφνικά ο κύριος Λάικιν να είναι στη Βαρσοβία, θα αποφασίσει ότι «α, δεν θέλω να συνεχίσω, σταματάω». Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και επί τη βάση των προτάσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαπιστώσετε ότι πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο τροπολογημένο νομικό πλαίσιο θα επηρεάσουν την σαφέστατη πλέον περιγραφή των αναγκών των επιχειρησιακών σχεδίων και της αξιολόγησης επίσης της δράσης του Frontex ένα στοιχείο το οποίο ίσως τα τελευταία χρόνια να μην ήταν ιδιαίτερα ισχυρό. Αυτά είχα να συμπληρώσω <clears throat> και να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι η ευθύνη των μεθοριακών φορών είναι ευθύνη του κράτους μέλους. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση την οποία θα έχουμε για μια πιθανή μελλοντική ε, ευρωπαϊκή μεθοριοφυλακή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα πάρα πολύ πρόωρο στάδιο και δεν θα πρέπει από την πρόταση αυτή να πιστέψει κανείς ότι θα υπάρξει μια μετάθεση ευθυνών προς την κοινοτική υπηρεσία. Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου έχει το λόγο. Θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. η ανταλλαγή απόψεων μου φάνηκε ιδιαίτερα καρποφόρος. Ελπίζω να επανέλθουμε για το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και στο Συμβούλιο. Πράγματι, ορισμένα κράτη-μέλη θέλουν την αρμοδιότητα να την έχει η Frontex όσον αφορά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, να μπορούν δηλαδή να το κάνουν αυτό. Φυσικά η πλαισίωση πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ καλή, να περιγραφεί πολύ καλά η αρμοδιότητα αυτή, να ξέρουμε πολύ καλά για ποια προσωπικά δεδομένα μιλάμε, ποια τέτοια δεδομένα μπορεί να έχει η Frontex, για ποιο στόχο και όλα αυτά τα κριτήρια και προϋποθέσεις να τηρούνται. Όλα αυτά ευθυγραμμίζονται απόλυτα με αυτά τα οποία εσείς είπατε σήμερα. Ε, προσπαθούμε να ετοιμάσουμε μία πρόταση για την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαρίστως την πρόταση αυτή μόλις την έχουμε να σας τη στείλουμε ώστε να ενημερωθείτε κι εσείς και έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Πρόεδρος, ο εισηγητής μας τώρα, ο κύριος Μπουσάτιλ, αλλά προηγουμένως να σας πω ότι προβλέπετε να παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής του εισηγητή στην επόμενη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. 13 Νοεμβρίου δηλαδή. Όχι, 15 διορθώνω ο πρόεδρος. 15, ε? Κύριε Μπουσούτιλ, τώρα έχετε το λόγο εσεί για τι τελευταίε παρατηρήσει επί του θέματο. Ευχαριστώ πολύ όλου του συναδέλφου που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε κάποιε διαφορέ σε μερικά σημεία, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να επιτευχθεί συνένεση για αυτό το ευαίσθητο θέμα. Κάποια σημεία θέλω να θίξω. Πρώτον, για την Ελλάδα. Φυσικά και με απασχολεί και εμένα πολύ και ανησυχώ για την κατάσταση στην Ελλάδα. Βέβαια το θετικό είναι ότι η Ελλάδα ζήτησε τώρα την ανάπτυξη δυνάμεων, πράγμα το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί η ρύθμιση. Και είναι μια πολύ κατάλληλη στιγμή αυτή, γιατί έτσι θα καταλάβουμε όλα αυτά τα οποία αποφασίσαμε το 2007 κατά πόσο αρκούν ή όχι. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να το διαπιστώσουμε αυτό. Η κυρία Ένστ ρωτάει τι ακριβώς θέλουμε από την Φροτεξ. Είναι η ερώτηση που παίρνει ένα εκατομμύριο δολάρια, έτσι. Κοιτάξτε, η συνθήκη επιτρέπει την αρμοδιότητα για τα εξωτερικά σύνορα να την έχουν τα κράτη-μέλη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι σε περιπτώσεις όπως είναι η Ελλάδα, όπου μία και μόνη χώρα νιώθει ότι έχει υπερβολικό φόρτο ή δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις μαζικές αυτές ροές λαθρομεταναστών, η Frontex είναι το καλύτερο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε όλες οι χώρες μαζί να πάνε και να βοηθήσουν τη μία εκείνη χώρα μέλος που έχει τη δυσκολία. Φυσικά η Frontex θα πρέπει να μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί τη αποστολή τη. Για την κυρία Βίλστρομ. Μίλησε για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και άλλοι συνάδελφοι. Σωστά είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την αρμοδιότητα να πει ναι ή όχι σε διακανονισμούς με τρίτες χώρες, αλλά λέει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται. Συμφωνώ μαζί της. Και όντω πρέπει να συμπεριλάβουμε κάτι εδώ, ώστε κάθε φορά που η Frontex κάνει διακανονισμούς για συνεργασία με τρίτες χώρες, εμείς να ενημερωνόμαστε. Η κυρία Γκυγιόμ τώρα είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για κάθε δραστηριότητα της Frontex. Αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο. Δηλαδή, πόσο μακριά θέλουμε να πάμε στο δημοκρατικό έλεγχο της υπηρεσίας αυτής. Πολύ βασικό το ερώτημα και θα προσπαθήσω με την βοήθειά της να το λύσουμε. Το Κοινοβούλιο θέλει δημοκρατικό έλεγχο πάνω στη Frontex για την επεξεργασία δεδομένων τώρα, προσωπικών δεδομένων. Όπως είπε κάποιος, θα βρεθούμε αύριο με την EDPS με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Υπηρεσία. Οπότε θα φροντίσουμε την αρμοδιότητα αυτή να την έχει η Frontex εφόσον, εφόσον, και το υπογραμμίζω, εφόσον έχουμε τις εγγύσεις που χρειάζονται ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά κάθε αυτά τώρα. Το έχω πει και άλλη φορά, αλλά το ξαναλέω. Όταν πήγαμε στην Βαρσοβία, το μήνα που μας πέρασε, και συζητήσαμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Frontex μας ξεκαθάρισε μέσω του Διευθυντή ότι η υπηρεσία έχει ανοχή μηδέν για οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πολύ χαρήκαμε που το ακούσαμε αυτό, γιατί δείχνει ότι η υπηρεσία δεν έχει κρυφή ατζέντα γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενισχύσει τις σχετικές διατυπώσεις στην ε, πρότασή της, οπότε πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με τους συναδέρφους, ώστε να φανεί ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υπάρχουν ισχυρέ διατάξει για την προσθέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλο, για την αγορά εξοπλισμού. Αναφέρθηκε σε αυτό η κυρία Βίξομ και η κυρία Γιόμ. Εδώ εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητήματα και οι ερωτήσεις ζητούν απάντηση. Κατά πόσο δηλαδή έχει νόημα να αγοράζει εξοπλισμό η υπηρεσία και ποιος θα ελέγχει τον εξοπλισμό αυτό. Ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να καταγράφει τις αγορές, ποιος θα δίνει οδηγίες για την αγορά τέτοιων εξοπλισμών. Αυτά είναι ζητήματα και προκύπτουν και νομικά ζητήματα πριν αποφασίσουμε θετικά. Τέλος, για το χρονοδιάγραμμα. όντω, στην επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα, ελπίζω να έχω έτοιμη την έκθεσή μου και έτσι να συζητήσουμε και για προθεσμία όσον αφορά την υποβολή τροπολογιών και για το πότε θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Ελπίζω και προσδοκώ ευρεία συνένεση πάνω σε αυτό το θέμα και για άλλη μια φορά ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους που με βοήθησαν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ποσότελ και την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη σημερινή συζήτηση. Θα ξανασυζητήσουμε για αυτό το τόσο λεπτό και το θέμα. 15 Νοεμβρίου, έτσι. Επί τη ευκαιρία της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής μας, της ΛΥΜΠΕ. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο πριν ε, το διάλειμμα. που προβλέπεται για τις 12.30. Τι έχουμε τώρα λοιπόν. Έχουμε ένα επιπλέον θέμα, το σημείο 12. Και αυτό είναι η καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Εδώ θα μας παρουσιαστεί μία μελέτη. Ξέρετε ότι όσον αφορά την κατάσταση πραγμάτων για το άσυλο, έχει γίνει μία μελέτη η οποία εξετάζει όχι μόνο την νομική πτυχή, δηλαδή τι ισχύει, αλλά κάνει και προτάσεις. Εξετάζει τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της νομοθεσίας. Οι συντάκτες της μελέτης αυτής όπως σας είπα, κάνουν και προτάσεις για το πώς μπορούμε να βοηθηθούμε στο κοινοβουλευτικό μας έργο. Ο κύριος Φίλιπ Ντεμπρέικερ, που είναι επικεφαλής του δικτύου, είναι εδώ στο Προεδρείο και θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αναλύσης αυτής. Και μετά θα έχουμε συζήτηση μεταξύ μας. Σας υπενθυμίζω όμως ότι η συζήτηση αυτή θα ακολουθηθεί από ερωτήσεις, μια μισή με τρεις, που μπορούν να υποβληθούν στην αίθουσα α1ε2. Εκεί θα είναι τα μέλη του δικτύου και μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις και θα μας απαντήσουν. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι εκεί. Έχει στελεί πρόσκληση στην ομάδα εργασίας για το άσυλο, αλλά όλοι οι ευρωβουλευτές μπορούν να πάνε εφόσον επιθυμούν. Α, άλλαξε η αίθουσα. Α5Ε2. Α5Ε2 είναι η αίθουσα. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Ντεμπρόικερ ευθύ αμέσω και μετά θα συζητήσουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει βέβαια πρώτα να σας ευχαριστήσω που μας δέχεστε σήμερα εδώ και να ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει με την ανάθεση της έκθεσης που ερχόμαστε σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Φυσικά, Πρέπει αμέσως να επισημάνω ότι μόνο μια σχηματική παρουσίαση της, ε, και λακωνική παρουσίαση της εκθέσεως μπορώ να πραγματοποιήσω, λόγω και του χρόνου που έχουμε στη θέση μας και του περιθωρίου να σας αφήσω, να αφήσω ένα περιθώριο για Ε, Μπορώ να μιλήσω λοιπόν για ένα 15 λεπτό και να παρουσιάσω μέσα σε αυτό μία έκθεση 500 σελίδων. Όπως καταλαβαίνετε θα είμαι πολύ λακωνικός και παρακαλώ οτιδήποτε δεν καλύψω, θετικό ή αρνητικό, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε θέση ή δεν έχουμε τίποτε να πούμε. Απλώς θα περιοριστώ στα ουσιοδέστερα. Τρία σημεία λοιπόν αποσχόλησαν την έκθεση κατόπιν τη του Κοινοβουλίου, του αιτήματο του Κοινοβουλίου, μα ζητήθηκε να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το κεκτημένο στο χώρο του, στον τομέα του ασύλου μπορεί να αξιολογηθεί. Ε, επισημαίνω εδώ ότι το πρόγραμμα της Χάγης απαιτούσε εν προκειμένου συστηματική, αποτελεσματική, αδέκαστη και αντικειμενική αξιολόγηση. Κατά την εξέταση λοιπόν των όσων έχουν γίνει και εν μέρει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι της αξιολόγησης των αιτήσεων, γιατί μπορεί να είναι ανεπαρκής αυτή, υπερβολικά νομική ίσως, και θέλω να επισημάνω επίση ότι στο επίπεδο το νομικό δεν έχουμε πάντω στη θέση μα τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία για να αξιολογήσουμε ε, μια αίτηση παραδείγματι πίνακε αντιστοιχία για τη μετάθεση στο εθνικό δίκαιο κάποιων οδηγιών ή των σχετικών διαταξιών του, των επιμέρου διαταξιών του. 50 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινοτικού Δικαίου Δυστυχώ ακόμη δεν έχουμε μπορέσει να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη ακριβεί πινάκες αντιστοιχεία σε Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο, πράγμα το οποίο σημαίνει μεγάλο χάσιμο χρόνο και για την Επιτροπή και για τους εμπειρογνώμονε. Ε, που χρειάζεται να δώσουν τις ε, πραγματογνωμοσύνες τους. Η αξιολόγηση πολλές φορές γίνεται κατακόρυφα μέσω συγκεκριμένων δηλαδή στοχεύσεων και όχι με οριζόντια μέσα ή γενικά μέσα. Επίσης επισημαίνεται ότι στο σύστημα του Δουβλίνου για τον προσδιορισμό του α, α, ε, υπευθύνου κράτους υπάρχουν ε, προβλήματα εφαρμογή και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεροληπτεί υπέρ τη διατήρηση του status quo, του φυσταμένου συστήματο, δηλαδή, του οποίου δεν θέλησε να αναθεωρήσει τι βασικέ αρχέ. Τώρα, υπάρχουν κάποιε πρόπτικε βελτίωση στο πεδίο αυτό. Ναι, μπορούμε και με τη βοήθεια του Γραφείου Στήριξης για τα θέματα του ασύλου που παρό, το γεγονός ότι θα είναι κατά πρώτο λόγο τουλάχιστον είναι σε πρώτη φάση αρμόδιο για να προσδιορίσει τι δικέ του αρμοδιότητε, αλλά θα μπορέσουμε να στηριχθούμε και στη δική του βοήθεια. Και με βάση νομική, το άρθρο 70 τη Συνθήκη Λισαβόνα, μια νέα νομική βάση για την αξιολόγηση των οδηγιών, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια προκειμένου, και παρά το γεγονό ότι, όπως θα έχετε κι εσείς ε, διαπιστώσει και κατά τρόπο παράλογο, έχει σχεδόν αποκλειστεί από την κοινοτική πολιτική του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με όλες λοιπόν τις επικρίσεις που μπορεί κάνει να διατυπώσει σε όλες αυτές τις μπορούμε νομίζω να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολη η αξιολόγηση, απαιτεί χρόνο μέσα και ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι, από ό,τι φαίνεται, διατεθειμένα ακόμη να στρατευτούν στην υπόθεση αυτή. Ε, μια ανακοίνωση της Επιτροπής ήδη το 2006 έκανε λόγο για τέτοια πράγματα, απερίφθη όμως από το Συμβούλιο ξεκάθαρα, γιατί θεωρούσε ότι είναι και πολύ... Ε, βαρύς, βαρύες οι δομές, αλλά και δαπανηρές, αυτά που πρότεινε δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά. Τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση του κεκτημένου και τις βραχυπρόθεσμες προτάσεις, τη δεύτερη φάση δηλαδή την οποία τώρα γνωρίζουμε και που στόχο έχει το, η θέσπιση ε, κοινού συστήματος ασύλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012. Έχουμε να κάνουμε πέντε ερωτήματα στα οποία θα ήθελα να αφαιρθώ. Πριν όμως, μια γενική παρατήρηση. Στην έκθεσή μας αξιολογούμε εν γέννη θετικά και μάλιστα θα έλεγα πολύ θετικά την πρόταση επαναδιατύπωση του συστήματο που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχε πάρει τον σωστό δρόμο και που σημαίνει ουσιαστικά ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλό θα κάνουν να ακολουθήσουν τι προτάσει τη Επιτροπή πλην μια ε, επιφύλαξη, την οποία ήδη ανέφερα, αλλά υπενθυμίζω, ότι πιστεύουμε ότι το σύστημα του Δουβλίνου θα έπρεπε να αναδιατυπωθεί. Είναι ανεπαρκής δηλαδή οι νέες ε, και κυρίως δεδομένε τη εξωτερική διάσταση του ασύλου που συνεπάγεται πολλές ανησυχίες, προβλήματα, έστω και αν αυτή η πτυχή δεν καλύπτεται τουλάχιστον 100% από τις προτάσεις που ε, δετυπώνονται για συζήτηση. Πέντε θέματα λοιπόν για την έκθεσή μας, καταρχάς το σύστημα του Δουβλίνου και η κατανομή των ετούντων το άσυλο και των προστατευνόμενων ατόμων. Το σύστημα του Δουβλίνου, το οποίο χαρακτηρίζεται από αδικίες ως προς τον ε, ετούντα το άσυλο και από ανισό, ε, ανισότιμη ε, επιβάρυνση των κρατών μελών, είναι ένα μη ε, ουδέτερο σύστημα, πράγμα το οποίο σημαίνει πολλά ε, μειονεκτήματα. Η δυνατότητα τώρα με την κατάθεση της ε, προσφυγής να εξασφαλιστεί αναστολή της, του επαναπατρισμού, της επανεισδοχής, ίσως μπορεί να αποτελέσει μια καλή λύση αφού δεν υπάρχει ικανοποιητική εξέταση της προσφυγής. Η αναστολή λοιπόν φαίνεται ότι ικανοποιητικά λειτουργεί, εκτός από κάποια τα οποία έχουν ε, ε, εξασφαλίσει ανασχετική μειονψηφία στο Συμβούλιο τουλάχιστον, αλλά πάντως η πρόταση είναι ευπρόσδεκτη, έστω και αν τη θεωρούμε ανεπαρκή. Πάντως θα πρέπει να απορριφθεί η απουσία αποτελεσματικότητα του συστήματο τώρα. Έχουν εντυπωθεί κάποιε προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα του συστήματο, αναθεώρηση των προθεσμιών, ε, διαδικασία ε, συνδιαλλαγή, συμφιλίωση. Ε, όμως δεν είναι επαρκείς αυτές οι προτάσεις, διότι δεν επιλύουν το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή την αδικία, το, το, μη ε, ισοδίκαιο σχηματισμό αυτού του συστήματο του Δουβλίνου, που επιβαρύνει ιδιαίτερα εκείνο τον ετούντο ο οποίο δεν θέλει να συνεργαστεί με το κράτο μέλο για, για να επιστρέψει στο κράτο από το οποίο έχει προέλθει. Ε, μια και δεν έχω πολύ χρόνο λοιπόν, δεν θα αναφερθώ στην οδηγία χαρακτηρισμού, μια και είναι το πιο ουδέτερο ζήτημα ουσιαστικά. Υπάρχουν κάποια επιμέρου σημεία μόνο, αλλά όχι επί της αρχής, για τον προσδιορισμό του ε, ατόμου ή του ποιος αναγνωρίζεται ως, ε, ως δικαιούχος του καθεστώτος της προστασίας ή της επικουρικής προστασίας. Πάντως δεν έχουμε ουσιαστικές ε, παρατηρήσεις για την οδηγία αυτή και την πρόσφυγη επιτροπής, η οποία όπως είπα μας φαίνεται καλή και σκόπιμη. Όσον αφορά τώρα το καθεστώ των προστατευμένων ατόμων και ιδιαίτερα τι συνθήκε υποδοχή των ετούνων το άσυλο, δύο είναι οι πτυχέ επί τη αρχή, τι οποίες ε, έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή, είναι η κράτηση, καταρχάς, και δεύτερον, ε, το ζήτημα των ευάλωτων προσώπων. Για την κράτηση των ετούνων το άσυλο, και πάλι ε, πολύ επιγραμματικά, έχει κάνει κάποιες προτάσεις αιτιών, μάλλον λόγων κράτηση η Επιτροπή. Το Συμβούλιο θέλει να διευρύνει τον κατάλογο αυτό, πράγμα που ε, εμεί δεν βρίσκουμε σκόπιμο. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εισαχθεί, με όλε τι δυσκολίε που μπορεί αυτό να σημάνει, μέγιστη διάρκεια κράτηση στην οδηγία για του ετούντε στο άσυλο. Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δηλαδή δεν μπορεί να επεφεθεί στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Χρειάζεται περισσότερη αναρμόνιση στο θέμα αυτό και επίση πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πως η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής ισχύει συγκεκριμένα στο σημείο στο οποίο κρατά, κρατείται ο ε, ετών το άσυλο, πράγμα το οποίο ακόμη εμφισβητείται. Για τις συνθήκες ε, υποδοχής. Το άτομο ο ετών το άσυλο ευάλωτης, ε, της κατηγορίας των ευάλωτων ε, ατόμων χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία. Εδώ λοιπόν και πολύ σωστά προβλέπεται από την οδηγία το ζήτημα του ποιος είναι αυτός ο οποίος θεωρείται ευάλωτος ε, και να δοθεί μια ειδική ρύθμιση που είχε ούτως ή άλλως ζητήσει η υφιστάμενη οδηγία, αλλά το κείμενο δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και ως εκ τούτου η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλά κάνει και κατατέθηκε. Πάντω φαίνεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, αλλά κυρίω του Συμβουλίου, προκύπτει ζήτημα ενοιολογικό και πλέον φαίνεται ότι δεν είναι πια σαφέ για το ποιον εννοούμε όταν μιλούμε για ετούντα το άσυλο ευάλωτο που έχει ιδιαίτερε ανάγκε κτλ. Εμεί θεωρούμε ότι είναι μία η έννοια. Ευάλωτο είναι το άτομο εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερε ανάγκε. Και επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους για να μην μπερδευτούμε. Επίσης, ε, σημειώνουμε πρόβλημα συντονισμού μεταξύ των κειμένων. Μια οριζόντια ανάλυση στην οποία επιδοθήκαμε δείχνει ότι χρειάζεται συντονισμό των κειμένων και της οδηγίας και των χαρακτηρισμών και του προσδιορισμού, του τρόπου προσδιορισμού των, ε, των ευάλωτων προσώπων. Επίσης, τίθεται ζήτημα που ίσως να μην μπορέσει όμως να επιληθεί εύκολα όταν γίνει ο προσδιορισμός, η ταυτοποίηση δηλαδή και ο τοπισμό των ευάλωτων προσώπων μέσα από όλες αυτές τις ε, ρυθμίσεις, μήπω θα ήταν σκόπιμο να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες ε, ταυτοποίησης των ετούντων το άσυλο υπό το πλαίσιο των συνθήκων ε, υποδοχής και μετά να υπάρχει μια άλλη οδηγία ε, για την εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου. Χωριστή δηλαδή διαδικασία που ενδεχομένως να σημαίνει περίπλοκες διαδικασίες και δυσκίνητες. Τέταρτον, όσον αφορά τις διαδικασίες για τη χορήγηση του ασύλου και πάλι θα είμαι όσο το δυνατόν πιο επιγραμματικός, βλέπουμε ως σημαντικό το γεγονός ότι η πρόταση αναδιατύπωση ενισχύει τι διαδικαστικέ, τι δικονομικέ δηλαδή εγγυήσει και πάνω απ' όλα σε ένα ε, νομικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται. Αυτό για εμά ως νομικού μα φαίνεται πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει να προσδιοριστούν τα όρια ή τα, ε, τα ορόσημα περισσότερο τη πολιτική ε, συζήτηση. Κάποια θέματα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν πολιτικά, διότι έχουν να κάνουν με νομικέ αρχές και δεσμεύσεις, δηλαδή το, δικαίωμα της προσωπικής προσφυγής, το δικαίωμα της προστασίας του προσώπου και μάλιστα όλα αυτά καλύπτονται από την ομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ή από την άλλη πρόκειται για κάποιες διατάξεις ε, συγκεκριμένες προστασίας των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι μπορεί η περιγραφή της, ε, του προβλήματος σχετικά φερειπίν με την δωρεάν παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, το ευεργέτημα της παινίας, να είναι ε, κάπως διαφορετική στην προκείμενη περίπτωση και να υπάρχει μια διαφορετική δυνατότητα λύση σε πολιτικό επίπεδο. Πέραν αυτού τώρα υπάρχει μια δυνατότητα εναρμόνισης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εναρμόνιση αυτού του τύπου των ε, διαδικασιών, την οποία και θεωρούμε ευπρόσδεκτη, αλλά φαίνεται ότι δεν μου φτάνει ο χρόνος μου για να επεκταθώ στο θέμα αυτό. Και θα περάσω στο πέμπτο σημείο, είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πρόθεσμα, θα έλεγα, είναι η εξωτερική διάσταση, μια εξωτερική διάσταση η οποία θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδης. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί, και αυτό είναι απόλυτα θεμητό, μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Έχουμε το σύστημα των θεωρήσεων, της κυρώσεις εις βάρος των μεταφορέων, την παρουσία συνδέσμων αξιωματικών για τη μετανάστευση και τα Frontex τις επεμβάσεις Frontex. Όλα αυτά τα μέτρα είναι θεμητά για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Ταυτόχρονα όμως μας φαίνεται και το επιβεβαιεί η Ένωση ότι θα παραμείνει ανοιχτή σε αυτούς οι οποίοι ζητούν άσυλο. Πάρα πολύ συχνά δεν μπορούμε να συνδυάσουμε με επιτυχία τις ανησυχίες μας από τη μία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του ανοίγματο προς αυτούς οι οποίοι θέλουν άσυλο. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα ε, του ασύλου είναι ένα θέμα το οποίο έχει υποβιβαστεί λίγο στις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται μέχρι τώρα. Στην ουσία φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αξιολογήσεις ή πολύ λίγες αξιολογήσεις των μέτρων τα οποία λαμβάνονται ε, για αυτούς οι οποίοι ζητούν άσυλο. Θα μπορούσε νομικά να πει κανείς βέβαια ότι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να γίνει επίκληση μάλλον αυτή της ευθύνη και υπερτοπικά δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον πρόκειται για κάτι το οποίο άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει λοιπόν η αρχή της μη επανέκδοσης Υπάρχει το δικαίωμα του ασύλου το οποίο αναγνωρίζεται πλέον στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το δικαίωμα σε αποτελεσματική και δίκαιη έφεση ε, ηλιμένων δικαστικών αποφάσεων. Τελειώνοντας, για να σεβαστώ ε, πάνω κάτω το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιο είναι το μέλλον του κοινού συστήματος χορήγησης ασύλου πέρα από τη δεύτερη φάση την οποία βιώνουμε και η οποία κανονικά τερματίζεται το 2012. Έξι προοπτικά μέτρα. Πρώτον, η νομική προοπτική. Είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο θα έλεγα υπάρχει στο ε, νομικό τοπίο, είναι η εγγραφή του δικαιώματος ασύλου στη χάρτα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πρόβλεψη αυτή είναι σημαντική αλλά και δύσκολη στην ερμηνεία της και ιδιαίτερα το θέμα της άμεσης, αν θέλετε, χρήσης του. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Υπάρχει μία ασάφεια για το πώς θα γίνει αντικείμενο ερμηνεία στο θέμα αυτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σχετικά τώρα με την ιδέα μίας ε, συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Σύμβαση της Γενέβης, όπως προβλέπει το πρόγραμμα της Στοκόλμης. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, αλλά θα υπάρξει ένα πρωτόκολλο ε, που τροπολογεί τη Σύμβαση της Γενέβης, όπως το κάναμε και με τη Σύμβαση για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, η ουσία δεν είναι να προσπαθήσουμε αν μπορούμε να το κάνουμε, είναι γιατί να το κάνουμε. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας συμμετοχής το ότι η Σύμβαση της Γενέβης επικυρωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην ουσία επιβεβαιεί τον ρόλο του κειμένου αναφοράς του συγκεκριμένου εγγράφου, της συγκεκριμένης συμβάσεως από πλευράς του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών διαφορετικό θέμα. Η δημιουργία ε, του γραφείου στήριξης ε, στους ετούντες άσυλο είναι επίσης κάτι το σημαντικό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απόλυτα έτοιμη να ε, διασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος αυτού στο μέλλον. Βλέπουμε ότι οι προτάσεις που γίνονται μέχρι τώρα λέγουν ότι οι υπηρεσίε αυτοί δεν έχουν καμία αρχή έμεση ή άμεση επί των εθνικών αρχών. Στην ουσία δηλαδή ε, εδώ έχουμε μια τροχοπέδη στην ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων και στην έβεθμη λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου. Ε, σε επίπεδο δικαιοδοσίας βλέπουμε ότι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην πολιτική ασύλου αυξάνεται συνεχώς μέσω των απαντήσεων που δίδει και μέσω των ερμηνειών που κάνει. Αυτό είναι θετικό. Είναι απαραίτητο αλλά είναι ανεπαρκές γιατί το δικαστήριο αποφασίζει επί δικαίου αλλά όχι επί πράγματι. Στην ουσία λοιπόν οι ε, καταστάσεις ε, παραμένουν πολλές φορές ακάλυπτες και δεν λύνουν τα προβλήματα. Νομίζω ότι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ασύλου δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό σε αυτή τη φάση. Η πρότασή μας λοιπόν για το μέλλον και εννοώ μακροπρόθεσμα είναι να φανταστούμε ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο για το Άσυλο θα μπορούσε να υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές, να τις αποστείλει στα κράτη-μέλη, με συνδρομή των δικαστών των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου, μέσω των ομάδων εργασίας, κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τα κράτη-μέλη, εφόσον βέβαια μπορούν να ερμηνευθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις. Αυτό υπάρχει σαν περίπτωση και στην πολιτική ανταγωνισμού, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατευθυντήριες γραμμές που έχουν, ε, θα έλεγα, αναγνωριστεί από την δικονομία και από τις αποφάσεις του δικαστηρίου που είναι πάντα παρόν για να επιβεβαιώσει την ε, ε, εγκυρότητα των κατευθυντηρίων γραμμών την εγκυρότητα της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών από τα κράτη-μέλη χωρίς να διαταραχθεί η συνταγματική τάξη. Τώρα, οι υλικέ προοπτικές. Ε, σας άκουσα να λέτε σήμερα το πρωί ότι στις περιπτώσεις ε, της χορήγησης αδείας μακράς διαρκείας ε, στους πρόσφυγες ε, είναι μια λύση η οποία δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική αν και σχετικά θετική. Νομίζω ότι μπορούμε εδώ να βρούμε ε, κάποιες ε, ομοιότητες με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή μετά την πρώτη ανανέωση της άδεια παραμονής να υπάρχει μια νέα τριετής περίοδος. Σχετικά τώρα με την ε, ε, διαδικασία κατανομής, το σύστημα Δουβλίνου δηλαδή. Το καθεστώς ακόμα και βελτιωμένο μέσω νέων προτάσεων δεν είναι βιώσιμο στο μέλλον και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσει του άρθρου 80 της συνθήκης που απαιτεί ότι η αλληλεγγύη θα πρέπει πρακτικά να λαμβάνεται υπόψη. Πρέπει να βρούμε διαφορετικά πρότυπα. Προτείνονται δύο πρότυπα. Το πρώτο πρότυπο είναι τη ύπα τη Αρμοστία και ε, το πρότυπο αυτό διατηρεί την αρχή της ευθύνη μεν, αλλά ε, ε, ιδιαίτερα για το κράτος το οποίο έχει γίνει συγκεκριμένη αίτηση εκτός από κάποιες εξαιρέσεις για οικογενειακούς λόγους. Το πρότυπο αυτό μας φαίνεται θετικό, είναι ένα πρότυπο το οποίο ε, πολλές φορές εξοικονομεί ε, μετακινήσεις σε περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης και ενώ το δεύτερο μοντέλο είναι το μοντέλο της ελεύθερης επιλογής, το οποίο μπορεί να είναι ιδανικό από πλευρά σε αυτών που ζητούν άσυλο, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό. Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με κλίδες κατανομής των ετούντων άσυλο ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι θέμα βέβαια υπολογισμών, μπορεί να υπάρξουν ποσοστώσεις στα κράτη-μέλη και όταν τα κράτη-μέλη φτάσουν σε μία ποσόστοση αλλά έχουν περισσότερες αιτήσει, τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να πάρουν μια αυξημένη βοήθεια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, να υπάρξουν και χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων μετακίνησης προσώπων που δεν θα ήταν στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, αλλά θα ήταν υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη, αλλά εθελοντικά για τους πρόσφυγες, γιατί πώς θα μπορούσε κανείς να φανταστεί την βίαιη μετακίνηση ετούν τον άσυλο. Τελειώνοντας, ε, θα ήθελα να περάσω στην εξωτερική προοπτική. Οι εξωτερικές προοπτικές έχουν γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων πρόσφατα, ιδιαίτερα μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου γύρω από το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η εξέταση των αιτήσεων ε, σε, στο πλοίο επάνω ε, δεν είναι κάτι το εφικτό, γιατί δεν δίδεται και η δυνατότητα έφεσης και νομίζω η προσφυγή, και ο καλύτερος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε κάποιες διαδικασίες προστατευμένης εισόδου όπως ακριβώς έχει προταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι τώρα από μία μελέτη η οποία δεν έγινε, δεν υπήρξε συνέχεια γύρω από αυτό. θα μπορούσε να υπάρξει μια θεώρηση περιορισμένης εδαφικής θα έλεγα ισχύως. Και θα πρέπει να βρούμε επίσης και ένα ουδέτερο στοιχείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με σφαιρικό τρόπο των μετακινήσεων πληθυσμών χωρίς να αγνοούμε τις διεθνείς πρόπτικες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά το θέμα της διεθνούς προστασίας ειδικά για το θέμα της διεθνούς προστασίας και να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εργαστούμε σε ένα ουδέτερο επίπεδο που πολλές φορές οδηγεί σε καλά αποτελέσματα σε επίπεδο διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και αναφέρομαι στη διάθεση της Χάγης στην οποία συμμετέχουν οι χώρες προορισμού αλλά και οι χώρες προέλευσης. Αυτό θα ήταν ένα κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαθέταμε περισσότερη ουδετερότητα και αντικειμενικότητα για τη συζήτηση ευαίσθητων θυμάτων λίγο περισσότερο από ένα τέταρτο πρόεδρε. Σας παρουσίασα με πολύ συνθετικό τρόπο τη μελέτη αυτή. Ελπίζω σήμερα το απόγευμα να έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε στη μελέτη των λεπτομεριών των συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία έθεσα και των συστάσεων τις οποίες κάναμε προσπαθώντας να σας δώσω την τελική έκθεση η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι το Μάιο του 10 και που περιλαμβάνει τις συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχετικά με την οδηγία υποδοχής και την αναμεταρρύθμιση της ε, συνθήκης του Δουβλίνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει προχωρήσει η ώρα, οπότε θα περάσουμε αμέσω στη συζήτηση που θα είναι όμω σύντομη. Ε? Η κυρία Γκάνα από πλευρά τη ε, Επιτροπή, παρακαλώ πρώτα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια νιώθει ήλιγκο με όλες αυτές τις ιδέες, τις τόσο ενδιαφέρουσες που ακούσαμε. Δεν συμμεριζόμαστε πάντα βέβαια την αξιολόγηση, αλλά πιστεύω ότι τέτοιες μελέτες ακαδημαϊκού χαρακτήρα και τόσο πλήρης μας βοηθούν να σκεφτούμε πολύ περισσότερο σε βάθος και να βρούμε πρακτικές λύσεις για να προχωρήσουμε και σε διαπραγματεύσεις αλλά και σε προβληματισμό όσον αφορά το ευρωπαϊκό κοινό καθεστώς ασύλου. Πολλές δυνατότητες δίνονται, σε όσα μας είπε ο Φιλίπ Ντεμπρέκερ, που αναφέρονται όμως ήδη στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, είτε πρόκειται για την εξωτερική διάσταση, είτε πρόκειται για τις διαδικασίες προστατευμένης εισόδου. Τέλος, συμφωνούμε απόλυτα με τους συντάκτες της μελέτης όσον αφορά τον πίνακα συσχετισμών. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μα ακόμα για τη συζήτηση. Ποιο είχε ζητήσει το λόγο, κάποιο είχε ζητήσει το λόγο. Κυρία Βέμπερ, πού είναι. Α, εκεί. Παρακαλώ, κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις είχα, αλλά νομίζω ότι απαντήθηκαν τελικά. Η μία ήταν να δούμε ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα Δουβλίνου, γιατί είπατε, αν σας κατάλαβα καλά, ότι ακόμα και τώρα όταν ξανασυζητάμε για το Δουβλίνο ε, δεν δουλεύει. Λοιπόν, ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να δουλέψει. Δεύτερον, είπατε ότι κάνατε μια οριζόντια αξιολόγηση των διαφόρων οδηγιών. Εδώστε μας μια ιδέα πώς μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο που βρισκόμαστε, όπου συναντάμε αντιφατικά ε, θέματα μέσα στην διαδικασία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ζίμπελ. Θα ήθελα και εγώ να είμαι σύντομη όσο μπορώ. Ένα από τα κύρια προβλήματα της, είναι αυτό της αλληλεγγύης των κρατών μελών όταν έχουμε δηλαδή ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν πολλά, πολλές ροές, πολλούς πρόσφυγες, τότε θα πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο δυνατό να διευκρινιστεί το ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος ε, αιτείται άσυλο και εκεί θα πρέπει ίσω να δοθεί κάποια υποστήριξη στα κράτη-μέλη και, πώς, και επίσης στο θέμα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών δώσετε κάποιες ποσοστώσεις, ίσως δεν είναι ξεκάθαρο, δώσετε κάποια, μιλήσετε για κάποιες ποσοστώσεις, ίσως δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι δεσμευτικές αυτές οι ποσοστώσεις. Και ίσως τελικά θα πρέπει η λύση να είναι να κατανέμονται κάπως αυτές οι αιτήσεις ασύλου μεταξύ των κρατών μελών. Για δε τα τρίτα κράτη. Ειδικότερα το ζήτημα της του ασφαλούς τρίτου κράτους. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, αξιολογείται το θέμα αυτό, τι είναι τρίτο κράτος, γιατί αύριο θα έχουμε και το θέμα της Λιβύης να συζητήσουμε. Εγώ προσωπικώς έχω σημαντικές επιφυλάξεις για το κατά πόσον ε, σε μια περίπτωση όπου η Λιβύη καθίσταται συμβαλόμενο μέρος ή προσπογράφει τη συνθήκη της ε, Γενέβης, δεν ξέρω αν αυτομάτως μετατρέπεται και σε ασφαλές τρίτο κράτος. Αυτό πώς το κρίνετε εσείς, ο κύριος Μπρόνς. Σύντομα. Τι αναλογία ετούντων άσυλο έρχονται κατευθείαν από τις χώρες από τις οποίες θέλουν να φύγουν και, από, και πόσοι έρχονται από ασφαλείς χώρες. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Thank you, Mr. Chairman, and I'd like to thank and congratulate the speaker for his uh, presentation. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, λέει ο κύριος Πουσότελ. Εγώ δεν ε, διάβασα, δεν είχα το χρόνο να διαβάσω ε, όλο το κείμενο, αλλά την παρουσίασή σας τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα και που μιλάτε για την αλληλεγγύη. Και είναι το λογικό συμπέρασμα αυτό στο οποίο καταλήγεται. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλη αντίσταση. Αλλά όπως και εσείς, έτσι και εγώ πιστεύω ότι αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάρουμε. Δύο θέματα θέλω να θίξω εγώ, πιο πρακτικής φύσεως. Θέλω όμως την άποψή σας. Πρώτον, ποια είναι η θεμητή πρόσβαση στο άσυλο, τι εννοώ δηλαδή. Έχει υπάρξει πίεση και εξακολουθεί να υπάρχει από την, άλλη μεριά θέλουμε, από την μια μεριά θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη λαθρομετανάστευση, από την άλλη μεριά θέλουμε να επιτρέψουμε στον κόσμο να έχει πρόσβαση στο άζυλο. Είναι μια συνεχής ένταση μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να καταπολεμούμε τη λαθρομετανάστευση και να στέλνουμε πίσω τον κόσμο από όπου και αν έρχεται και άλλοι πολύ σωστά λένε ότι αν το κάνουμε αυτό τότε παραβιάζουμε την αρχή της μη επιστροφής όντως υπάρχει μια παράνομη δραστηριότητα που αν την επιτρέπουμε γινόμαστε συνένοχοι. Αν δείτε την αντοχή μηδέν ε, δεν είναι μυστικό για κανέναν ποιοι οργανώνουν τις μετακινήσεις αυτές. Αν λοιπόν επιτρέψουμε ε, το άσυλο μέσα από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες γινόμαστε συνένοχοι με την εγκληματικότητα. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, υπάρχουν πραγματικοί τρόποι μέσω των οποίων να μπορούμε να προσφέρουμε το άσυλο, αλλά με νόμιμο τρόπο και όχι να βοηθάμε τις εγκληματικές διαδικασίες. Αυτό είναι το ένα. Επίτα. πρέπει να ξέρουμε ότι το κόστος είναι τεράστιο και ότι είναι δύσκολο να πουλήσουμε εντό αγωγικών αυτά που λέμε σε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει βρεθεί για αρκετό καιρό μάλιστα σε δύσκολη κατάσταση. Και τι λέμε στην Ελλάδα, τις λέμε ότι και δεν τα καταφέρνεις να τα βγάλεις πέρα και να τηρήσεις ε, την κατάσταση σε ανεκτά επίπεδα, αλλά ε, Κάνει και μεγαλύτερε παραβιάσεις ακόμα. Λοιπόν και για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες που βρίσκονται στην Νότια Ευρώπη τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό θα ήθελα τη δικιά σας αντίδραση, να μου πείτε τη γνώμη σας. Πώς μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, ποιε λύσεις μας προτείνετε για τέτοιε δύσκολε καταστάσει που αντιμετωπίζουν ορισμένε χώρες μέλη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κανένα άλλο που θέλει το λόγο. Α, ο κύριο Σταβάρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Ντεμπρόκερ, για την παρουσίασή σα που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και γεμάτη πληροφορίε. Έχω μια ερώτηση, έμεση κάπως, όσον αφορά το θέμα της επανακατάστασης. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε εγκρίνει δύο σχετικές εκθέσεις, μία ιδίας πρωτοβουλίας και μία άλλη με συναπόφαση. Σε εκείνη ιδίας πρωτοβουλία. είπαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μία μονάδα επανεγκατάστασης με το κατάλληλο προσωπικό. 10-15 δεν είπαμε τον αριθμό, αλλά κάποιοι που να δουλεύουν γι' αυτό. Για μετανάστες. Πώς επανακατίστανται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. έχουμε σκεφτεί πού θα μπορούσε να κατασταθεί αυτή η μονάδα και είπαμε σε άτυπο διάλογο που είχαμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι ίσως το γραφείο για το άσυλο να είναι ο καλύτερος χώρος για να κατασταθεί η μονάδα αυτή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, πιστεύετε κι εσείς ότι θα ήταν καλό ένα άλλο κομματάκι της διαχείρισης και της κάλυψης όλων αυτών των φαινομένων όντως να τοποθετηθεί εκεί στο άσυλο. Και να γίνεται έτσι και η σύνδεση με άλλες υπηρεσίες, την και κλπ. που δουλεύουν για τους πρόσφυγες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες. Ο χρόνος περνάει. Δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Οπότε, ο κύριος Δεμπρέκη παρακαλώ να απαντήσετε Πάρα πολύ σύντομο όμως, γιατί έχουμε περάσει το χρόνο μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα με υποχρεώσει η οδηγία σας να είμαι πολύ πιο συνοπτικός από ότι ήμουνα υπερβολικά θα έλεγα. Πρώτον για το Δουβλίνο και τη λειτουργία του Δουβλίνου. Νομίζουμε ότι το Δουβλίνο δεν μπορεί να λειτουργήσει για μια ολόκληρη σειρά από λόγους. Πρέπει να επανεξεταστεί το σύστημα είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη φάση για να αξιολογήσουμε ουσιαστικά τη λειτουργία του συστήματος και το αναβάλαμε για μια ακόμη φορά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακριβώς κάποιες αρχές του συστήματος του Δουβλίνου, το ότι δεν μπορεί κανείς παρά να κάνει μία φορά αίτηση και στη χώρα άφηξης κτλ. είναι κάποιες αρχές θετικές, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν τα συστήματα μεταφοράς, τα οποία έτσι και αλλιώ είναι περιορισμένα. Τα περισσότερα από αυτά δεν ε, λειτουργούν ουσιαστικά και κοστίζουν πάρα πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το σύστημα του Δουβλίνου έτσι και αλλιώς γενικότερα. Δεύτερον, σχετικά με την οριζόντια αντιμετώπιση του θέματος ανάμεσα στις ε, πολλαπλές οδηγίες. Δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι ε, να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν βλέπω άλλη λύση. Νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει μια κάποια προσπάθεια εκεί όπου υπάρχει ανάγκη συντονισμού, υπάρχει ένα θέμα το οποίο τίθεται συνεχώς, είναι το θέμα του ορισμού των μελών της οικογένειας, ποια είναι μέλη της οικογένειας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι τόσο σημαντικό το θέμα και μπορεί να, τόσο δύσκολο μάλλον και μπορεί να δοθεί απάντηση. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Μπορούμε να βασιστούμε στο άρθρο 80 της συνθήκης για να πούμε ότι από εδώ και πέρα η οργάνωση της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν είναι θέμα πολιτικό. Είναι μια υποχρέωση νομική την οποία θα πρέπει να οργανώσουμε σωστά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ξεκαθαρίζεται. Τώρα για ποιες είναι ασφαλείς χώρες. Αυτό που μου φαίνεται περίεργο είναι ότι στα πλαίσια της οδηγίας στα πλαίσια της νέας σύνταξης ε, καταργείται ε, ο καθορισμός του καταλόγου ε, ευρωπαϊκού και να παραπέμπουμε μόνο σε εθνικούς καταλόγους. Έτσι κι αλλιώ έχουμε αμφιβολίες για τη χρησιμότητα αυτής της έννοιας, γιατί έτσι κι αλλιώ υπάρχουν πολλές λειτουργικές απαιτήσεις για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών, τα οποία έτσι χάνουν τις δυνατότητες που έχουν για γρήγορη και σωστή εξέταση της περίπτωσης σχετικά με τις ροές. Δεν είμαι ικανός να απαντήσω για το αν έρχονται απευθείας από τη χώρα τους ή περνούν από κάποιες άλλες χώρες διαμετακόμισης. Αυτό δεν ήταν στόχος της μελέτη μας. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που έχουν στατιστικά στοιχεία στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπα, τη αυμοστία δεν θα ήταν σε θέση να δώσουν μια ουσιαστική απάντηση. Τώρα για την ερώτηση του κυρίου Μπουσούτιλ για τις μικτές ροές. Πράγματι εδώ η προβληματική τίθεται και με πολύ απαιτητικό τρόπο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί υπάρχει ένα παράδοξο το οποίο γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα στα πλαίσια του οποίου επενδύουμε πολύ σε ενέργεια και δεν ε, προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό το πολυτελές σύστημα μπορεί να γίνει αντικείμενο πρόσβασης από τους ενδιαφερομένους. Υπάρχει παράδοξο εδώ λοιπόν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε το δικαίωμα αναζήτησης του ασύλου με την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Είναι νομική συζήτηση, είναι περίπλοκη συζήτηση, υπάρχει το θέμα της υπερτοπικής ευθύνης, υπάρχει το θέμα της ερμηνείας του δικαιώματος στο άσυλο. Όλα αυτά είναι δύσκολα νομικά θέματα. Υπάρχουν όμως και ορισμένες ε, ιδεοντολογικές διαστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παραμείνει εν μια ανοιχτή ήπειρος και φοβάμαι ότι πολλές φορές ε, απεκδιόμεθα τις ευθύνη την οποία έχουμε, κάτι το οποίο νομικά μπορεί να είναι τεκμηριωμένο αλλά πολιτικά είναι κάτι το οποίο δεν προστατεύει αυτούς που έχουν δικαίωμα στην προστασία αυτή. Λοιπόν, το θέμα του δικαιώματος ασύλου και του κόστους του είναι πολιτικό περισσότερο, παρανομικό. Και πράγματι οι προτάσεις βελτίωσης οι οποίες γίνονται έχουν ένα κάποιο κόστος. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με αυτό, σε σχέση με την κατανομή των πόρων, με τη διάρκεια των διαδικασιών, αν θα πρέπει να βραχύνουμε τις διαδικασίες, αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να αποφύγουμε διαδικασίες οι οποίες κρατούν πάρα πολύ και να προσπαθήσουμε να τις καταστήσουμε πιο γρήγορες. Και στο τέλος, για την επανεγκατάσταση και για την υπηρεσία βοήθειας και συνδρομής, ναι και πάλι ναι, εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να στηρίξουμε, χρειάζεται χρόνος έτσι ώστε να πείσουμε για την ανάγκη αυτής της δημιουργίας ε, ε, της υπηρεσίας αυτής στήριξης. Χάσαμε πολύ χρόνο σε επίπεδο πρακτικής συνεργασίας γιατί δεν υπήρχε καθοδηγητική ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι το γραφείο αυτό θα προχωρήσει. Είμαστε πεπισμένοι ότι στην ουσία θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε και όχι τόσο ε, στο μέλλον τις δυνατότητες διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του γραφείου αυτού, γιατί αυτή είναι η πορεία του μέλλοντος. Εν πάση περιπτώσει δεχτήκαμε να το, να το δημιουργήσουμε. Είναι ένα θετικό βήμα. Βέβαια του στερούμε πολλές δυνατότητες. Είναι λυπηρό το να γράφουμε ότι η υπηρεσία αυτή δεν έχει καμία αρμοδιότητα, έστω και έμεση σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Σαν να μην θέλαμε να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που αποφασίσαμε να ανοίξουμε. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι αυτή είναι η γραμμή που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια, όχι αύριο, αλλά σε 5-10 χρόνια. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διακόπτουμε εδώ. Και θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα στην ίδια αίθουσα για να συνεχιστεί η συγκεκριμένη συνάντηση στις 3. Ευχαριστώ και την διερμηνία για τον επιπλέον χρόνο. Ο